Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς ένα μήνυμα από τους διερμηνείς. Είναι η 36η ημέρα της διαμαρτυρίας μας κατά της μονομελούς επιβολής ανισόρροπων και άδικων συνθήκων εργασία για του διερμηνεί από πλευρά τη διοίκηση του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λυπούμαστε λοιπόν, που σα ενημερώνουμε ότι η διερμηνία θα ε, σταματήσει στην προγραμματισμένη ώρα λήξη τη συνεδρίαση. Σα ευχαριστούμε για την κατανόησή σα. Όπως είχαμε αποφασίσει ε, στους συντονιστές θα ακούσουμε την παρουσίαση της μελέτης από το Ίδρυμα Ανοιχτή Κοινωνία ε, για τα πορίσματα τη σε ό,τι αφορά την κατάσταση των μουσουλμάνων γυναικών στην Ευρώπη. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μαριά Χμαντούν από του ε, συγγραφεί τη μελέτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Μάλιν Μπιόρκ κυρίω ε, για την πρόσκληση, γιατί χρειάζεται πραγματικά γενναιότητα και θάρρο για να θέσουμε ένα τέτοιο ζήτημα στη, στο παρόν πολιτικό κλίμα της Ευρώπης είναι πολλά τα διακυβευόμενα και καλό θα είναι να αντιληφθούμε ότι οι φεμινιστές, οι φεμινίστριες από όπου και προέρχονται θα πρέπει να συσπυρώσουν τις δυνάμεις τους, να δημιουργήσουν μια συμμαχία για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ανακύπτουν. Και γι' αυτό θέλω να είμαστε υπέρ μια πιο δίκαιης, ανοιχτής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. so before I... Πριν ε, σας παρουσιάσω τα απορίσματα μιας ε, μελέτης και έκθεσης που εκπονήσαμε, θα ήθελα να σας εξηγήσω τι ακριβώς κάναμε και για ποιο λόγο. Του χρόνου, το 2019 δηλαδή, στη Γερμανία, ε, η κοινωνία των πολιτών και κυρίως πολλές μουσουλμάνες γυναίκες θα Έχουμε την επέτειο του θανάτου της Μαρουέλ Σαρμπίνη, της πρώτης γυναίκας ε, που φορούσε μαντίλα και ακριβώς σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε για αυτό το γεγονός, επειδή ήταν μουσουλμάνα που φορούσε μαντίλα. Ε, και πάλι είχαμε μία επίθεση ε, κατά μίας μουσουλμάνας ε, πρόσφατα, πριν από μία εβδομάδα, μόνο και μόνο επειδή φορούσε μαντίλα. Πριν από 10 χρόνια λοιπόν είχαμε τη δολοφονία μιας γυναίκας ε, μουσουλμάνας επειδή φορούσε μαντήλα, αλλά έχουμε και συνεχείς επιθέσεις ε, ε, προς μουσουλμάνες, είτε τις έφτυναν, τις τραβούσαν τις μαντήλες, είτε τις που πετούσαν μπουκάλια μπύρας, υπέστησαν πολλές σωματικές επιθέσεις και μάλιστα η έκθεση μας δεν αφορά αυτά τα εγκλήματα μίσους, σεξιστικά και μισαλόδοξα εις βάρος των μουσουλμάνων και κυρίως των μουσουλμάνων ε, γυναικών. Οι γυναίκες οι μουσουλμάνες ε, φαίνεται ότι ε, μερικές φορές νιώθουν να μην έχουν θέση σε αυτήν την κοινωνία. Η έκθεση μας όμως δεν φορά αυτά τα εγκλήματα μίσους, αλλά τα διαρθρωτικά προβλήματα που οδήγησαν σε τέτοια κατάσταση. Και συζητήσαμε κάποιες πολιτικές και νομοθετικές διατάξεις που θεσμοθετήθηκαν και που χαρακτηρίζονται από αυτή την ε, στιγματιστική εμπριστική ρητορική βάρος των μουσουλμάνων γυναικών που ουσιαστικά δικαιολογούνται τις επιθέσεις. Ε, η έκθεση έγινε σε 20 χώρες μέλη, αφορά μάλλον την κατάσταση για πολλές χώρες μέλη. Χαρτογραφεί όλους τους περιορισμούς που δικαιολογούνται από τις ίδιες μορφές ε, καταστολής και καταπίεσης ε, ναι. των μουσουλμάνων γυναικών, τον αποκλεισμό τους από την απασχόληση, την παιδεία ή το δημόσιο χώρο. Όλους αυτούς τους τομείς καλύπτουμε στη μελέτη μας. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι τομείς στους οποίους οι μουσουλμάνες γυναίκες υφίστανται διακρίσεις, αλλά αυτή είναι η βασική τομής. Οπότε οι κανόνες αυτές όχι μόνο δημιουργήσαν φραγμούς στη μελετη μας φυσικα υπαρχουν και αλλοι τομει στους οποιους οι μουσουλμανες γυναικες υφιστανται διακρισεις αλλα αυτη ειναι η βασικη τομη οποτε οι κανονες αυτες οχι μονο δημιουργησαν φραγμους στη συμμετοχη στον οικονομικό, κοινωνικό και δημόσιο βίο για τις γυναίκες μουσουλμάνες, αλλά ποινικοποίησαν ουσιαστικά την παρουσία τους, την προβολή τους, την ίδια τους την ύπαρξη στην κοινωνία μας. Οπότε η σύνταξη της σχετικής έκθεσης ήταν πολύ σημαντική για μας γιατί ένας πολίτης αξιοπρεπής θα ήταν κατά τέτοιων εγκλημάτων μίσους σίγουρα ε, η αγανάκτηση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη αν η κατάσταση ήταν διαφορετική. Αν δηλαδή λευκές ε, γυναίκες, μη μουσουλμάνες ήταν τα θύματα σε επιθέσεις από μουσουλμάνους. Οπότε ε, μπορεί να υπάρχει απόρριψη για τέτοια εγκλήματα, αλλά δεν υπάρχει τέτοια απόρριψη των νομοθετικών διατάξεων που οδηγούν ή δημιουργούνται υπόβαθρο για αυτά τα εγκλήματα, για αυτές τις συμπεριφορές. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να έχουμε μια πιο ανοιχτή, ανεκτική κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς. Και παρά την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι το αποτέλεσμα τέτοιων νομοθετικών μερικέ φορέ περιορισμών ή πολιτικών και που έχει αναγνωριστεί από όλα τα δικαστήρια και παρόλο που αποδυναμώνεται και φέρει σε δυσμενή θέση μια ομάδα γυναικών που ούτω ή άλλω υφίστανται ε, διακρίσει λόγω ε, τη θρησκεία ή της εθνότητάς τους ε, παρόλο βέβαια που πολλές έχουν γεννηθεί και ανατραφεί στην Ευρώπη, υφίστανται τις ίδιες ε, διακρίσεις ε, λόγω φύλου, αλλά έχουν επιπλέον περιορισμούς επειδή φαίνεται ότι είναι μουσουλμάνες γυναίκες. Και κανονικά έχουν το δικαίωμα εξηθρησκεία και δεν το απολαμβάνουν όμω ούτε την ελευθερία έκφραση και ελευθερία συνείδηση. Και επιπλέον έχουν μια οικονομική εξάρτηση. Κάτι που εμποδίζει τη χειραφέτησή του. Γιατί, γιατί ε, επικρίνονται για την επιλογή του ενδυματολογικού τους κώδικα, που είναι έκφραση της ε, πεποίθησης ότι πρέπει να καταπιέζονται, ότι δεν μπορούν να σκεφτούν από μόνες τους, ε, ότι δίνουν νόημα στο τι σημαίνουν τα ρούχα τους, τα ενδύματά τους και ότι δεν μπορούν να πρωτοστατούν στην προάσπιση των δικαιωμάτων των δικών τους ή γενικώ των δικαιωμάτων των γυναικών. Κάνουμε μια κρίση λοιπόν λόγω του, της ενδυματολογικής επιλογής και την επεκτείνουμε σε μια συμπεριφορά. Κρίνουμε τι γυναίκε από τα ρούχα του και από το νόημα που δίνουμε σε αυτά τα ρούχα και μάλιστα τι τιμωρούμε για αυτήν την ενδυματολογική του επιλογή. Και νομίζω ότι αυτό είναι από τα πιο παλιά πατριαρχικά, φαλοκρατικά τεχνάσματα. Ότι οι γυναίκε ε, δεν δίνονται μόνο με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά ειδικά οι μουσουλμάνε δίνονται με συγκεκριμένο τρόπο. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια αντίφαση. Θα πίστευε κανεί ε, ότι γι' αυτό το λόγο απειλούν την κοινωνία μα. Ο τρόπο που ντύνονται, ε, όχι μόνο δείχνει την άγνοια του στην αδημοσύνη του, αλλά είναι ταυτόχρονα ε, απειλή για την κοινωνία μα. Υπονομεύει τι ε, αξίε μα. Και αν τι αποδεχτούμε θα υπονομεύσουν ό,τι πιστεύουμε, όλε τι αρχέ και τι αξίε μα. Άρα, μουσουλμάνε γυναίκε σημαίνουν απειλή. Αυτό που κάνουμε λοιπόν στην έκθεση είναι να χαρτογραφήσουμε όλου αυτού του περιορισμού που είναι κυρίω εξιστικοί και ρατσιστικοί περιορισμοί. Και σε πολλές χώρες οι περιορισμοί αυτοί δημιούργησαν ένα ολόκληρο ιστό ένα ευρύτατο δίκτυο περιορίζοντας υπερβολικά τις ε, μουσουλμάνες γυναίκες ε, και στην ε, άσκηση της θρησκείας τους και τη συμμετοχή στο δημόσιο ή επαγγελματικό βίο. Μερικές φορές οι γυναίκες αυτές δύσκολα εμφανίζονται ε, δημοσίως χωρίς να γίνονται θύματα επιθέσεων. Συνέχως προσκρούν σε τέτοιους περιορισμούς. Βλέπουμε λοιπόν ποια είναι τα προβλήματα, ποιε είναι οι βασικές νομοθετικές προτάσεις αλλά βλέπουμε και κάποια, κάποιο θεσμικό υπόβαθρο, δηλαδή τους κανονισμούς που έχουν εγκριθεί είτε καταστατικά από σχολεία, <laughs> από ιδρύματα, από ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, και ε, έχουν σημαντικό αποτέλεσμα. Επίσης, είδαμε πολιτικές πλατφόρμες και πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν σε τέτοιους περιορισμούς σε διάφορες χώρες, προσπαθώντας να αντιληφθούμε ταυτόχρονα την αιτιολόγηση που δόθηκε για να υιοθετηθούν τέτοιοι νομοθετικοί περιορισμοί και γενικώ την ρητορική που του συνόδευσε. Τα συμπεράσματά μας είναι τα εξή. Αυτό είναι ένας χάρτης των περιορισμών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Και διαπιστώσαμε ότι συνολικά εννέα χώρες έχουν νομικού περιορισμού για του θρησκευτικού ενδυματολογικού κώδικες ε, με της μουσουλμάνες γυναίκες, με στόχο τις μουσουλμάνες γυναίκες. Βλέπετε ε, το κόκκινο. Οι χώρες με κόκκινο έχουν εθνικούς περιορισμούς. Η Γαλλία είναι η χώρα με τους περισσότερους ε, και πιο ευρύς ε, περιορισμούς και πιο μακροχρόνιους περιορισμούς. Υπάρχει εθνική απαγόρευση για το πέπλο προσώπου, ε, για τα, τις μαντήλες στα σχολεία και στους επαγγελματικούς χώρους. Η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Δανία έχουν, απαγορεύουν επίση το πέπλο προσώπου. Μερικέ χώρε έχουν μερικού περιορισμούς που εφαρμόζονται εθνικά. Για παράδειγμα, έχουμε μία απαγόρευση μόνο σε συγκεκριμένου τομεί, όπως πρόσφατα είχαμε κάτω χώρε. Εθνικό μεν περιορισμό που περιορίζεται όμω σε συγκεκριμένου τομεί. Στην υγεία, στι δημόσιε συγκοινωνίε και ούτω καθεξής. Επίση, έχουμε κάποιε άλλε χώρε, Γερμανία για παράδειγμα, Ιταλία, Ισπανία και Βέλγιο πάλι, που έχουν κάποιους τοπικούς περιορισμούς, περιορισμούς δηλαδή που είναι μεν νομικοί, αλλά ισχύουν σε συγκεκριμένες περιοχές ή πόλεις. Οπότε βλέπετε τις χώρες που έχουν θεσμοθετήσει κάποιους νομικούς περιορισμούς. 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάποιους θεσμικούς περιορισμούς. Δηλαδή Έχουμε σχολεί συγκεκριμένε επιχειρήσει που έχουν υιοθετήσει τέτοιου περιορισμού, που περιορίζουν την πρόσβαση δηλαδή στι μουσουλμάνε γυναίκε. Ε, και επίση σε πέντε χώρε συζητούν αυτή τη στιγμή νομοσχέδια. Ε, το Βέλγιο ήδη έχει κάποιου περιορισμού ε, και συζητά περαιτέρω περιορισμού, ενώ νομοσχέδια συζητούν και άλλε χώρε που δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει τέτοιου περιορισμού ενδυματολογικού για τι μουσουλμάνες. 14 χώρες αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζουν περιορισμούς. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί από τις 22 χώρες που εξετάσαμε, ε, στις περισσότερες χώρες ε, συζητήθηκαν κάποια στιγμή νομοσχέδια που όμως απορρίφθηκαν. Αυτό είναι θετικό. Δηλαδή, ναι, με κατατέθηκαν νομοθετικέ προτάσει, αλλά απορρίφθηκαν. Και σε 22 χώρε ε, έγιναν νομοθετικέ συζητήσει για τέτοιου είδου μέτρα. Και διαπιστώσαμε ότι αυτή η όθηση, αυτή η πρόταση για τη νομική έγκριση τέτοιων περιορισμών αυξάνεται. Υπάρχει μια τέτοια αύξουσα τάση, ανωδική πορεία για τη θεσμοθέτηση περιορισμών. Μάλιστα, η έκθεση εκπονήθηκε τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, δύο επιπλέον χώρε ε, θέσπισαν ή ενίσχυσαν του νομικού περιορισμού. Και μάλιστα σε μια χώρα είχαμε περισσότερη νομολογία για τέτοιου κανονισμού που απαγορεύουν τη μαντήλα στα σχολεία. Επίσης, κάποιες χώρες είπαν ότι προτίθενται να προτείνουν νέε νομοθετικές προτάσεις. Οπότε υπάρχει μια τέτοια νοδική τάση για τέτοιους περιορισμούς. Και μάλιστα έξι χώρες μόνο ουδέποτε δεν συζήτησαν πρόταση για περιορισμό. Μόλις τώρα έχουν υποβληθεί κάποιες προτάσεις με την ανάλυση των συμπερασμάτων ε, καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι οι νομικοί περιορισμοί είναι σχετικά μικρής ε, εμβέλειας ευτυχώς, αλλά μέσα σε λίγους μήνες είχαμε δύο νέους ε, νομικούς περιορισμούς για θρησκευτικά ενδύματα. Επίσης, με την ανάλυση των διαφόρων επιχειρημάτων και την εξέλιξη αυτών των περιορισμών στις διάφορες χώρες, βλέπουμε ότι η άκρα δεξιά και τα εθνικιστικά κόμματα ζητούν περισσότερους περιορισμούς πιο ε, εξαπλωμένους, πιο ευρύς και διαδεδομένους. Και παρά, τη σχετικά ζωφερή και απεσιόδοξη κατάσταση, αυτό που με εμψύχωσε κάπως και μου έδωσε ελπίδες, είναι ότι οι κυβερνήσεις, τα εθνικά δικαστήρια και τα διάφορα ιδρύματα κάπως υπαναχώρησαν σε ό,τι αφορά την αρνητική του στάση απέναντι στι μουσουλμάνες. Για παράδειγμα, έχουμε κάποια δικαστήρια που απέρριψαν τη θεσμοθέτηση περιορισμών στο παρελθόν σε χώρε όπω η Γαλλία και το Βέλγιο που έχουν πολυάριθμους περιορισμού. Και οι μουσουλμάνες φαίνεται ότι ενεργοποιούνται και δραστηριοποιούνται στην κοινωνία των πολιτών καταρρύπτοντας τέτοιε πολιτικέ. Επίση, έχουμε ιδρύματα και επιχειρήσει που προωθούν πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς που έχουν βρει τρόπο να ε, επιτρέψουν και να καταστήσουν δυνατή την ισότιμη συμμετοχή των διαφόρων ομάδων, ε, ανάλο, άσχετα με το ηθονοτικό, θρησκευτικό ή άλλο υπόβαθρό τους. Οπότε είναι σαφές ότι παρά τις προσπάθειες επικρατεί μια πολύ αρνητική ρητορική εις βάρος των μουσουλμάνων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, των γυναικών κυρίως. Και παρά το γεγονός ότι πολλά εθνικά δικαστήρια απέρριψαν τους περιορισμούς ε, σε θρησκευτικούς ειδηματολογικούς κώδικες ε, ε, δεν βρήκαν αρκετές αποδείξεις για να καταρρύψουν τα ναι. επιχειρήματα υπέρ των, περιορισ... των περιορισμών. Και δυστυχώς, ενώ τα εθνικά δικαστήρια είναι πιο αρνητικά κατά των περιορισμών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο προστατεύονται αυτές οι αποφάσεις. Στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουμε πολλές τέτοιες υποθέσεις και έχουμε μία εξέλιξη της νομολογίας. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση για το τι συμβαίνει επί τόπου. Μέχρι στιγμής πάντως τα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν ήταν τόσο προστατευτικά όσο τα εθνικά δικαστήρια για τις μουσουλμάνες. <coughs> και φτάνω στα συμπεράσματα Ποια συμπεράσματα μπορούμε να αντλήσουμε από την ανάλυση μας. Υπάρχουν αδιάστητες αποδείξεις ότι οι περιορισμοί στρέφονται κατά των μουσουλμάνων γυναικών. Και αυτοί, αυτές οι απαγορεύσεις, ε, όταν είναι τμήμα πολιτικών ή ε, νομοθετικών διατάξεων, είναι γενική κάπως και όριστη. Πάντως η βάση, ε, η αιτία αυτών των περιορισμών και η αρχική τους διατύπωση πολύ συχνά ε, οι αρχικοί νομικοί περιορισμοί στρέφονταν αρχικά κατά της μαντήλας. Μετά αποφάσισαν να έχουν μια πιο γενική διατύπωση για να μην κατηγορηθούν για διακρίσεις βάρος των μουσουλμάνων. Οπότε έγιναν πιο εκλεπτισμένες οι διατυπώσεις, πιο γενικές, γιατί εμείς παρόλα αυτά γνωρίζουμε ότι στόχος αυτών των περιορισμών είναι οι μουσουλμάνες. Θέλουν τον αποκλεισμό των μουσουλμάνων. Αυτές είναι στο στόχαστρο όλων αυτών των πολιτικών. Και πολύ συχνά σε πολλές χώρες υπήρχαν και εξαιρέσεις για άλλες εκφάνσεις ε, ε, άλλων θρησκειών, της καθολικής, της ε, εβραϊκής. Για τέτοιες θρησκείς υπήρχαν εξαιρέσεις, ενώ για τους μουσουλμάνους όχι. Όλα αυτά είναι αποδείξεις ότι όλοι αυτοί οι κανόνες στόχο είχαν να αποκλείσουν τις μουσουλμάνες. Και όλοι το γνωρίζαμε, αλλά τώρα έχουμε αποδείξεις που στηρίζουν αυτή τη θέση. Και φυσικά δεν θα ερχόμασταν εδώ να σας μιλήσουμε αν δεν πιστεύαμε ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ειδικά η Επιτροπή σας, ε, ε, μπορούν να κάνουν κάτι για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Μπορείτε να μας βοηθήσετε, ε, να αναγνωρίσετε δημοσίως και να πείτε ότι αυτός ο αποκλεισμός των μουσουλμάνων μέσω των περιορισμών στον ενδυματολογικό του κώδικα είναι και σεξιστικός και ρατσιστικός. Γιατί να μην υποβάλλετε προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ρωτώντας πώς συμβιβάζεται αυτή τη, αυτόν τον αποκλεισμό των μουσουλμάνων με τις αρχές της ισότητας των φύλων και το, τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουμε κάνει διαβήματα προς διάφορους φορείς και όργανα για να εξεταστούν τα αποτελέσματα που έχουν τέτοιοι νομικοί περιορισμοί ε, για τα ενδυματολογικά στις μουσουλμάνες και πώς επηρεάζουν γενικώ την πρόσβασή τους. Γιατί με τέτοιες προσπάθειες θα βοηθήσουμε να απελευθερωθούν οι γυναίκες, να χειραφετηθούν και να σταματήσουν οι καταπιέσεις και οι καταστολές. Γιατί όταν δούμε τι αποτέλεσμα έχουν αυτοί οι περιορισμοί στι μουσουλμάνε, βλέπετε ότι όχι μόνο δεν τι χειραφετούν, όχι μόνο δεν τι απελευθερώνουν, αλλά τι κάνουν και το βίο αβίωτο. Γιατί προσάρμοσαν τι επιλογέ του και τη ζωή του ε, στην ελεύθερη άσκηση της θρησκείας τους. Θέλαμε λοιπόν οι διάφοροι φορείς να διερευνήσουν τι συμβαίνει επί τόπου, γιατί χρειαζόμαστε τέτοια στοιχεία και τέτοιες αποδείξεις για να τεκμηρώσουμε τις αγωγέ μας ε, στα δικαστήρια, γιατί φαίνεται ότι τα δικαστήρια δεν έχουν επαφή με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και επίση, να διοργανωθούν και δημόσιες ακροασει, να καλέσετε ε, ως μάρτυρες αυτές τι γυναίκες για να σας μιλήσουν για του περιορισμού που υφίστανται. Επίσης, ε, θα πρέπει να προωθήσουμε μια ανοιχτή κοινωνία, χωρί αποκλεισμού. Γιατί γνωρίζουμε την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δέχτηκε με κάποια μορφή πολλούς περιορισμούς και κυρίως την απαγόρευση κάποιων ε, ενδυματολογικών συμβόλων. Και αυτό σίγουρα στρέφεται εις βάρος μιας ανοιχτής κοινωνίας ε, και ενισχύει τους αποκλεισμούς. Ε, μιλάμε για τα δικαιώματα του ΛΟΑΔΜ. Αν αρκούσε μία δικαστική απόφαση για να ανοίξουμε την κοινωνία απέναντι στι εθνοτικέ και θρησκευτικέ μειονότητε στην Ευρώπη, δεν θα είχαμε όλα αυτά τα κινήματα ΛΟΑΔΜ, όλα τα αντιρατσιστικά κινήματα. Δεν θα χρειάζονται να αρκούσε μία δικαστική απόφαση για να ανατραπεί η νομοθετική πορεία. Χρειαζόμαστε περισσότερα από μία απόφαση δικαστηρίου. Γιατί πολλοί πολίτε αγνοούν την κατάσταση. Πρέπει εσεί να μα βοηθήσετε να προβάλλετε αυτέ τι αποδείξεις, τα τεκμήρια, να ρωτήσετε νομικούς εμπειρογνώμονες και να ε, δείτε γιατί αυτή η δικαστική απόφαση ναι μεν ε, υπάρχει, αλλά δεν αποκαθιστά τη δικαιοσύνη για τις γυναίκες αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να μας βοηθήσετε για να αποκατασταθεί αυτή η κατάσταση, να απονεμηθεί πραγματικά δικαιοσύνη στις μουσουλμάνες και η κοινωνία να γίνει πιο ανοιχτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την προσοχή σας. Thank Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαριάμ Μπακαντούλ, για αυτή την παρουσίαση της καταστάσεως που αφορά τις μουσουλμάνες γυναίκες στην Ευρώπη. Θα ακούσουμε ευρωβουλευτές τώρα. Και κυρία Βιόρκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ που ήρθες Μυρία να παρουσιάσει την έκθεση. Για μένα ήταν η πρώτη που διάβασα που έκανε γενική επισκόπηση των 28 χωρών. Σημαντικότατο να προχωρήσει η κατανόησή μας. Για να ξεκινήσω λοιπόν, θέλω να πω ότι το θέμα εντάσσεται στο ότι οι μουσουλμάνες γυναίκες έχουν προβλήματα στον αυτά τα δικαιώματά τους, τους επιτίθενται ακροδεξιές ομάδες, τις έχουμε και στο κοινοβούλιο αυτές τις ομάδες, όπως ξέρετε, υπάρχει μια, ε, αναφέρεστε στην κουλτούρα την ευρωπαϊκή που προσπαθούμε να έχουμε μια ενωμένη Ευρώπη. Η ακροδεξιά δεν το δέχεται. Δεν δέχεται ότι μπορούμε να ενωθούμε στη διαφορετικότητά μας και ότι μπορούμε να είμαι πλουραλιστική η κοινωνία μας. Αυτό είναι ένα κομμάτι της εικόνας. Οι συνάδελφοι της Επιτροπής πολεμάμε για την ισότητα των φίλων, τα δικαιώματα των γυναικών σε όλα τα πεδία, τα δικαιώματα όλων των γυναικών. Βέβαια, οι πάλι σας είναι και δική μας πάλι, αλλά πρέπει να μάθουν περισσότερα. Και κάποια από τους συναδέλφους εδώ θα θέλουν να μάθουν τις νομικές διεξόδους που υπάρχουν, πολιτικές δυνατότητες, τοπικές απαγορεύσεις, εθνικές απαγορεύσεις, γενικές απαγορεύσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη γενικότερη εικόνα, για τα νομικά ζητήματα. Πολύ ενδιαφέρουσα η άποψη, αυτά που μας είπες. Αυτή πάλι περνάει και από δικαστικές υποθέσεις, όπως και με κάθε πάλι χρειάζεται χρόνο. Έχει μια επιρροή η δικαστική απόφαση, χρειάζεται χρόνο για να επιδράσει. Πρέπει να είμαστε προσεκτικέ, να κινηθούμε προσεκτικά προ σωστή κατεύθυνση. Καμιά φορά έχουμε και ήττε, αλλά συνεργαζόμενε θα κινηθούν προ τη σωστή κατεύθυνση. Όταν το ΔΕΚ έλαβε απόφαση περί βγήκε μας ανησύχησε διότι δεν μας ικανοποιούσε αυτή η απόφαση. Χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια. Αυτό που είναι ενθαρρυντικό είναι ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Οι προτάσεις που έκανες για κοινοβουλευτικό ρώτημα στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα το κάνουμε είτε ως Επιτροπή, θα το συζητήσουμε αυτό βέβαια, είτε να παρουσιαστούμε σαν ομάδα μελών. Όποιος θέλει να συνεργαστεί μαζί μου, ας έρθει να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες, να το ερευνήσουμε το θέμα. Είναι καλό να λάβει ρόλο η κοινωνία των πολιτών, αλλά πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Να διοργανώσουμε ακροάσεις, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα που σε καλέσαμε, αλλά ίσω και σε μια κρόση θα μπορούσαμε να ακούσουμε και νομικούς και να μάθουμε και δικαστικές υποθέσεις. Υποσχεθήκαμε ότι θα είμαστε εταίροι προστατεύοντας τα δικαιώματα των γυναικών, των μουσουλμάνων γυναικών και θέλουμε κοινωνία που θα είναι ελεύθερη από κάθε μορφή διάκριση. Δεν θέλουμε να ζήσουμε σε μια σεξιστική και ρατσιστική κοινωνία. Ευχαριστώ. Η κυρία Πιτικάινεν. Δύο λεπτά σας παρακαλώ για ερώτηση-αντίδραση. Διότι έχουμε πολλή δουλειά. Πολλά θέματα. Κυρία Πιτικάινεν έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Κάποια σχόλια. Ίσως μπορούμε να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για να υποβάλουμε ψήφισμα στην Ολομέλεια ή να υποβάλουμε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα ως γνωστόν. προστατεύονται από τη διακήρυξη περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από διάφορα συνταγματικά δικαιώματα. Ποιο είναι το σημαντικό γεγονό. Πολλέ μελέτες δείχνουν ότι όταν κινδυνεύουν κοινωνίες και η δημοκρατία εν γέννη, πάντα οι γυναίκες και οι μειονότητες καταπιέζονται. Είναι γενικότερο θέμα από ότι το καναρίνι στο ρηχείο που δείχνει ότι λείπει το οξυγόνο ότι, υπάρχουν επιθέσεις από την άκρα δεξιά τώρα στην Ευρώπη. Έχουμε μάθει πράγματα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πώς ξεκινάνε αυτά. Όταν αρχίσουν οι αλληλοκατηγορίες και κάποιοι θεωρούν ότι άλλοι είναι λιγότερο σημαντικοί σαν άνθρωποι και έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους άλλους. Ελπίζω ότι μπορούμε σαν Επιτροπή να αντιδράσουμε από αυτού. Ίσως μαζί με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών σε εσάς να Η κυρία Μορβάη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική ευκαιρία όταν εμείς οι γυναίκες μπορούμε να συνομιλούμε σε ένα περιβάλλον αδελφών και να είμαστε ειλικρινεί. Με κάθε ειλικρίνεια η ερώτησή μας. Γιατί οι μουσουλμάνες γυναίκες θέλουν να φύγουν από τις κοινότητές τους σε επεκτεταμένες οικογένειές τους τα χωριά τους, τις παραδόσεις τους, τη θρησκεία τους κλπ. Να τα αφήσουν όλα αυτά πίσω, να έρθουν στην Ευρώπη. Και είτε να προσπαθήσουν να ζήσουν την ευρωπαϊκή του ζωή, είτε όπως είπατε εσείς, να κάνουν την Ευρώπη μουσουλμανική ή να κάνουν δικές κοινότητες και να ζήσουν μουσουλμανική ζωή. Αυτή είναι μια βασική σημαντική ερώτηση. Παρόλο που είστε πολύ πολιτισμένοι γυναίκα και εργάζεστε για την πρωτοβουλία ανοιχτή κοινωνία στην Ευρώπη και είστε πολύ μορφωμένοι. Ίσως όμως να έχετε και κάποια πιο βαθιά σχέση με τις αδελφές σας. Πείτε μας, για ποιο, ποιο είναι το κίνητρο. Υπάρχουν παράδοση, γλώσσα θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες. Αυτό το στηρίζουμε οι φεμινίστριες, διαδίδονται από γενιά σε γενιά. Γιατί να κόψετε τις ρίζες σας και να έρθετε στην Ευρώπη. Άλλη ερώτηση. Δεν είναι πάνω από δύο λεπτά και δεν υπάρχουν και μέλη. Οποιοςδήποτε μπορεί να καθίσει στην αίθουσα. Όλοι οι ψηφοφόροι βλέπουν ότι υπάρχουν ελάχιστοι βουλευτές. Έχουμε χρόνο Καταλαβαίνω ότι είναι ευαίσθητο το θέμα, αλλά παρακαλώ απαντήστε στην ερώτηση αυτή που είναι ευαίσθητη. Όλοι αυτοί οι άντρε καταφθάνουν. Άντρε, άντρε καταφθάνουν. Τι γίνεται. Οι μητέρε του, οι αδελφέ του, τι γίνονται. Οι γυναίκε του που μένουν πίσω. Και περιμένω την απάντησή σα. <coughs> Ευχαριστώ. Κυρία Κρουσίνσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δηλώσατε ότι οι επιθέσεις κατά των μουσουλμάνων γυναικών είχαν μικρότερη αντίδραση από ότι όταν δέχεται μια επίθεση από έγχρωμο άντρα μια λευκή γυναίκα. Λοιπόν, μετα... Στο... στην κολονία έγινε η επίθεση χριστουγεννιάτικα στην κολονία από μουσουλμάνους άντρες σεξουαλική βία και δεν είδα κάποια αντίδραση στο κοινοβούλιο. Θεωρείτε ότι είναι κάποια μορφή ελευθερίας το να φοράτε τη μαντήλα η πλειοψηφία των γυναικών στη, στη Γαλλία είναι υποχρεωμένε σε κάποιε κοινωνίε να καλύπτονται πλήρω ή να φορέσουν μαντήλα, αλλιώ δεν έχουν την άδεια να βγουν από το σπίτι του. Αυτό είναι η έννοια ελευθερία για εσά. Αντίθετα, οι γυναίκε, είτε είναι μουσουλμάνε ή όχι, δεν μπορούν να περπατήσουν σε κάποιε γειτονιέ στη Γαλλία πια χωρί να παρενοχλούνται ή να προσβάλλονται, ακόμα χειρότερα, και καμιά φορά δεν έχουν το δικαίωμα ε, να μπουν καν στα μαγαζιά. Και αυτή είναι η έννοια της ελευθερίας για σας. Καταγγείλατε τους εθνικούς νόμους, τις νομοθεσίες στην Γαλλία, κυρίως τα εμφανή σημάδια της θρησκεία. Εμεί το αποκαλούμε κοσμικότητα. Μέχρι τώρα το σύστημα λειτουργούσε αρκετά καλά. Αλλά με τις δικές σας πολιτικές διεκδικήσεις αυτή η κοσμικότητα έχει την τάση τελικά να κλονίζεται. Ευχαριστώ. η κυρία Μαριά μου να δώσει κάποιες απαντήσεις, παρακαλώ. Να απαντήσω καταρχάς στην πρώτη ερώτηση. Καταρχάς, να διασκεδάσω τις προϋποθέσεις σε πολλές από τις ερωτήσεις σας που δεν έχουν καμία βάση κατά τη γνώμη μου. Ε, μιλάτε για τις μουσουλμάνες γυναίκες, ε, λέτε ότι έρχονται από το εξωτερικό για να εξισλαμίσουν την Ευρώπη. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, δεν θέλουμε η Ευρώπη να γίνει μουσουλμανική. Η πλειοψηφία των γυναικών για τις οποίες μιλάμε γεννήθηκαν, μεγάλωσαν εδώ, εδώ είναι η πατρίδα τους ε, και στην κοινωνία της Ευρώπης θέλουν να συμβάλλουν. Στην Ευρώπη θέλουν να πάνε σχολείο, να συμβάλλουν οικονομικά, κοινωνικά. Εδώ θέλουν να έρχονται σε επαφή με τους συμπολίτες τους. Οι γυναίκες αυτές ε, συχνά έχουν υιοθετήσει και μιλούν τις πολλές γλώσσες της Ευρώπης δεν θέλουν να επιβάλλουν τη γλώσσα τους ή τις παραδόσεις τους. Θέλουν μόνο να απολάβουν των ίδιων δικαιωμάτων με τους συμπολίτες τους. Δεν ήρθαν εδώ, εδώ γεννήθηκαν. Δεν σκόπευαν ούτε σκοπεύουν να αλλάξουν τους κανόνες. Θέλουν να παραμείνουν οι κανόνες οι ίδιοι. Αυτά είναι τροποποιήσεις στο νόμο που έγιναν πριν κάποια χρόνια, το πολύ πριν μια δεκαετία, ε, σε χώρες όπως είναι η Γαλλία. Έγιναν τροποποίησεις στην νομοθεσία για να αποκλειστούν αυτές οι γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές θέλουν να παραμείνει η ίδια η νομοθεσία για να συμμετάσχουν επίσης όρις με άλλες γυναίκες. Δεν θέλουν να βλάψουν κανέναν δεν θέλουν ε, να αποτελέσουν κίνδυνο για κανέναν, θέλουν απλά να έχουν τα ίδια δικαιώματα και να ζουν με τον ίδιο τρόπο με γυναίκες μη μουσουλμάνες ή χωρίς ε, συγκεκριμένο ε, εθνοτικό υπόβαθρο. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, ως φεμινίστρια, ως γυναίκα που υπερασπίζομαι τα δικαιώματα των γυναικών καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου, είμαι κατά κάθε μορφής καταπίεσης και μαζί με όλες τις γυναίκες που αγωνίζονται για το θέμα αυτό, είμαστε εξίσου κατά της επιβολής της μαντήλας στις γυναίκες, όπως είμαστε κατά και της απαγόρευσης της μαντήλας. Θέλουμε οι γυναίκες μόνες τους να αποφασίζουν πώς ε, θα ε, ασκούν τη θρησκεία τους, τι θα φοράνε, εάν θέλουν να είναι θρήσκες ή όχι. Αυτό θα πρέπει να εναπόκειται στις γυναίκες. Μπορούν να σκεφτούν μόνες τους, μπορούν να λαμβάνουν μόνες τους αποφάσεις, να αποφασίσουν πώς θα ζήσουν τη ζωή τους. Αυτό εκτιμούμε στις χώρες στις οποίες ζούμε. Και είχαμε τις ελευθερίες αυτές. Θέλουμε να υπάρχει ισότητα για όλους. Πώς να γίνει αυτό μέσω των ίδιων θεσμών που οικοδομήθηκαν τα τελευταία χρόνια για να προστατεύσουν τις γυναίκες από τον ε, καταναγκασμό και την καταπίεση. Υπάρχουν κανόνες για να προστατεύσουμε τις γυναίκες αυτές. Ας ε, χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα, να μην ε, υιοθετούμε νέα νομοθεσία για να τις τιμωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Το να θεωρούμε ότι είναι όλες καταπιεσμένες θεωρώντας ότι είναι όλες καταπιεσμένες, τις τιμωρούμε όλες. Δεν βοηθάτε τις γυναίκες που φοράνε αναγκαστικά ε, ε, τη, τη συγκεκριμένη τη μαντήλα για λόγους θρησκευτικού. Ε, δεν θα πρέπει να με τιμωρείτε επειδή έχω την εμφάνιση που έχω και επειδή φοράω μαντήλα, ούτε να υποθέτετε ότι στηρίζω τέτοιου είδους καταπίεση. Ε, η λαϊσίτε, η κοσμικότητα που έχει μεταφερθεί και στις γειτονικές χώρες ως ουδετερότητα, πιστεύουμε ότι είναι πολύτιμη αρχή, διότι προστατεύει τα δικαιώματα όλων μας. Να πιστεύουμε ότι πιστεύουμε και να συμμετέχουμε στην κοινωνία. Στην ανάλυση αυτή τη έκθεση υπάρχουν όμω ακόμα και καλύτερε αναλύσει όπω του ε, Γάλλου Ζαμποτέρο δείχνει ότι η εφαρμογή της αρχής αυτής έχει αλλάξει σε βάθος χρόνου για να αποκλείσει τη συγκεκριμένη ομάδα από την κοινωνία. Είναι λοιπόν σημαντική αρχή. Και όπως η ισότητα των δύο φύλων, όπως η ανεξιθρησκεία, έχει χρησιμοποιηθεί η αρχή αυτή για να αποκλείσει μια συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. Και πιστεύουμε ότι αυτό υπονομεύει τις αξίες της Ευρώπης και τα ιδανικά που θέλει να πετύχει. Θέλουμε να πούμε ότι είναι δυνατόν και να έχουμε τις αξίες αυτές και να συμμετέχουμε στην κοινωνία. Δεν υπάρχει αντίθεση εδώ. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ. Thank you. Thank you very, Thank you for your presentation. Thank you for your answers. Ευχαριστούμε κυρία Μαρία Μουχαμεντούν για την παρουσίαση της έκθεσης και τις απαντήσεις σας. Σίγουρα πολλά έχουμε να κάνουμε και γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούμε. Now, uh, now the nine on agenda care services e Περνάμε στο σημείο 9. Υπηρεσίες παροχής φροντίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για βελτιωμένη ισότητα των φύλων. Το λόγο έχει η συγκεκριά μας, η κυρία Σιέρπα Πιετικάινεν. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, δεν θα σταθώ σε όλες τις λεπτομέρειες, θα σας παρουσιάσω μόνο τα βασικά σημεία. Καταρχήν υπάρχει διαχωρισμός στην κοινωνία μας, όπως γνωρίζετε. Και γι' αυτό ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο την κοινωνική διάσταση, αλλά την έμφυλη διάσταση και τη σκοπιά των γυναικών. Σίγουρα ε, πολλοί χρειάζονται φροντίδα και κυρίως στο σπίτι και 75% των παρόχων φροντίδα είναι γυναίκες. Και αυτό προκαλεί και δυσκολίες ε, στην επαγγελματική ζωή, στη σταδιοδρομία, στο επίπεδο αμοιβών, αλλά και στις συντάξεις που λαμβάνουν οι γυναίκες. Και στις κοινωνίες μας χάνουμε περίπου 370 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο λόγω της χαμηλής αμοιβή των γυναικών ή τις ανάγκες τους να παραμείνουν στο σπίτι ούτε καταφέρουν να συνδυάσουν καλά τον επαγγελματικό με τον προσωπικό τους βίο. Και αυτά τα προβλήματα θα οξυνθούν στο μέτρο που γυράσκει ο πληθυσμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν <laughs> μια τριπλή ε, βελτίωση. Καταρχήν χρειαζόμαστε καλύτερε υπηρεσίε υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και καλύτερη ποιότητα και καλύτερη πρόσβαση, αλλά και πιο προσιτέ τιμέ. Και κυρίω για το γεράσκοντα πληθυσμό θέλουμε φροντίδα ώστε ε, οι χρήζοντες φροντίδα να μπορούν να, ε, να την λάβουν είτε στο σπίτι τους κατοικών είτε στα συγκεκριμένα κέντρα είτε σε ε, νοσοκομεία, αλλά η πλειοψηφία α, α, και αυτών των των φροντίδα θα είναι γυναίκες, γιατί έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής. Επίσης, ε, υπάρχουν προβλήματα στι υπηρεσίε υγεία δυστυχώ ε, στην Ευρώπη και υγειονομική περίθαλψη. Οπότε θα πρέπει να βελτιώσουμε την παροχή υπηρεσιών υγεία και κάτι τέτοιο να ληφθεί υπόψη και στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ο δεύτερο πυλώνα ε, στη λύση του προβλήματο είναι τα εργασιακά δικαιώματα. Και οι γυναίκες όταν λαμβάνουν άδειε για να παράσχουν φροντίδα, θα πρέπει να ε, ισχύει κάτι παράλληλο με αυτό της ε, ε μητρότητας. Να υπάρχει δηλαδή δυνατότητα είτε άδεια μεταποδοχών, πλήρων αποδοχών, είτε μερικών αποδοχών. Και να υπάρχει δυνατότητα τέτοια χορήγησης άδειας για παροχή φροντίδας αλλά και άλλα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και υπάρχει μια πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους παρέχοντες φροντίδα. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι πάροχοι φροντίδας, να αναγνωρίσουμε την κατάστασή τους και να αντιλήσουμε κάποια συμπεράσματα και σε ό,τι αφορά τα εργασικά τους δικαιώματα και στα δικαιώματα αμοιβή, αλλά και στα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Θέλουμε επίσης υπηρεσίες παροχής φροντίδας, αλλά και υπηρεσίες στήριξης των παρόχων τη φροντίδα. Επίσης, θέλουμε οικονομική υποστήριξη για όσους αφιερώνονται στην παροχή φροντίδας. Και επίσης να προσφέρουμε υπηρεσίες και αποκατάσταση και φροντίδα στους παρέχοντες φροντίδα. Τέτοιου είδους υπηρεσίες προτείνουμε λοιπόν στο πρόγραμμα αναγνωρίζεται η αξιέπαινη έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά επίσης αναγνωρίζουμε και τις ε, προσπάθειες που θα πρέπει να γίνουν στο μέλλον. Ελπίζουμε η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναβαθμίσει το σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους παρόχους ε, φροντίδα. Αναφέρονται και οι δικές μας εκθέσεις, γίνονται Πολλέ μνήες των δικών μα προτάσεων, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που εγκύπτουμε στο θέμα αυτό. Επανειλημμένω έχουμε ασχοληθεί με το ζήτημα. Αυτά περιμένω τα σχόλιά σα και τι απορίε σα αν υπάρχουν. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Πιετικάινεν. Περνάμε στου και οδησηγητές και οδησηγήτριε. Η Μαρία Καβριέλα Ζωανά είναι η πρώτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγήτριά μας, την κυρία Πιέτε για τις παρατηρήσεις του. Για τις παρατηρήσεις Θέλουμε καλύτερες ε, παροχές φροντίδας και ε, βρεφικής και ηλικιωμένων. 38% των γυναικών ε, ασχολούνται με την ανατροφή των παιδιών τους, των εγγονιών τους ή ηλικιωμένων ή αναπηρών και αφιερώνουν τουλάχιστον μία ώρα τη μέρα σε τέτοια φροντίδα. Σε... Το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι 25%. 25%. Και σίγουρα οι τέτοιε ευθύνες, οι ευθύνε παροχή φροντίδας που έχει η γυναίκα οδηγεί στην λιγότερη πρόσβασή τη στην αγορά εργασία και στην ε, χαμηλή τη αμοιβή. Υπάρχουν λοιπόν με μεγάλες μισθολογικές διακρίσεις και μεγαλύτερος κίνδυνος στο γυναικό και κοινωνικό αποκλεισμό. Συμφωνώ με την εισηγήτρια και την έκθεση ότι οι υπηρεσίες φροντίδας θα πρέπει να αναπτυχθούν ε, περαιτέρω ώστε να ανταποκρίνονται στις ε, ανάγκες ανδρών και γυναικών και στην καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Επίσης θα πρέπει να ενισχυθούν οι παροχές ε, υπηρεσίες σε βρεφική παιδική ηλικία αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια ζωής και επίσης να δούμε πόσο προσιτές είναι οι τιμές, τι προσβασιμότητα υπάρχει και σε μακροπρόθεσμες υπηρεσίες φροντίδας και θα πρέπει να έχουμε κοινούς ορισμούς, καλύτερη συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη δικτών και στόχων. Επίσης, ε, έχω κάποια στοιχεία που θα υποβάλω με τις τροπολογίες μου. Γενικώ ε, θεωρώ ότι κάποιοι με χρόνιες παθήσεις χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα. Τέτοιου είδους ε, υπηρεσιών μακροχρόνιας παροχής φροντίδας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται. Επίσης, η ποιότητα τέτοιων υπηρεσιών φροντίδας και σε παιδιά και σε μακροχρόνια χρήζοντες θα είναι πολυδιάστατο φαινόμενο. Θα πρέπει να περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης, κοινωνικά, βελτίωση των υπηρεσιών, γιατί η ποιότητα των υπηρεσιών συνδέεται αναπόσπαστα με την ποιότητα ζωής των παρόχων φροντίδα. Θα πρέπει λοιπόν να τα εξετάσουμε όλα αυτά σε ε, επίπεδο εκπαιδευτικό αλλά και επίπεδο εργασιακών συνθήκων του προσωπικού που παρέχει φροντίδα. Σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα, η πληροφορία για τη διαθεσιμότητα τέτοιων υπηρεσιών φροντίδας θα πρέπει ε, να είναι ε, προσιτή και να ενημερώνεται και για την δυνατότητα επαγγελματική ανάπτυξης. 80% ε, ε, παροχής φροντίδας γίνεται από ανεπίσημους ε, παρόχους φροντίδας και κυρίως από γυναίκες. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε και κάποιο είδους σταδιοδρομία, επαγγελματική διέξοδο για την παροχή φροντίδας και όχι μόνο την άτυπη παροχή φροντίδας. Και έτσι θα έχουμε μεγαλύτερη παροχή ε, εκπροσώπηση των γυναικών και γι' αυτό θα πρέπει να ε, δώσουμε μεγαλύτερη επαγγελματική και ψυχολογική στήριξη στις γυναίκες για να εξασφαλίσουμε την, τον συνδυασμό επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Και χαίρομαι για την πρόταση σύσταση του Συμβουλίου για ε, καλύτερα συστήματα παροχής φροντίδας ε, και σε επίπεδο προσχολικής ηλικίας. Επίσης, ε, ζητούμε από τα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν τα τοπικά και εθνικά τους σχέδια με βάση τις συστάσεις και ζητούμε από τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα για να βελτιώσουν ε, την κατάσταση του τομέα ε, παροχής φροντίδας και να εξασφαλίσει την ε, ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων στην αγορά εργασίας. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της υπαίθρου, για παράδειγμα, ή τα παιδιά σε οικογένειες μεταναστών. Οι πολιτικές και τα προγράμματα στα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ε, καλύτερη πρόσβαση των μειονεκτούντων σε ε, υψηλών προδιαγραφών και των υπηρεσιών υγείας. Επίσης, να καταπολεμήσουμε την παιδική φτώχεια από τα πρώιμα στάδια της και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να ενισχύσει την υποστήριξή της σε άτομα ε, με μειονεκτικό υπόβαθρο και τα σχόλια μου αυτά θα τα συμπεριλάβω και σε τροπολογίες και προσβλέπω σε καλύτερη συνεργασία με την εισηγήτρια και τους άλλους ηγέτες για το θέμα αυτό. Η κυρία Κούνεβα έχει το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου την συνάδελφο Σύρπα Πιετικάινεν για το σχέδιο έκθεσης που μας παρουσιάζει σήμερα. Πριν ξεκινήσω όμως, θέλω να επισημάνω κάτι επί το διαδικαστικού. Δυστυχώς και αυτή την έκθεση έχει πέσει θύμα του θλιβερού ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ποιο έχει τη αρμοδιότητα. Το είδαμε στην επιστολή των συντονιστών της Επιτροπής Επασχόλησης που μας εστάλει. Το αποτέλεσμα είναι να στριμώχνονται χρονικά κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή σημαντικά κείμενα και ψηφίσματα που αφορούν εκατομμύρια πολιτών που εκπροσωπούμε. Είναι πολύ κακό σημάδι ότι δέκα μήνες πριν τις επόμενες ευρωεκλογές έχουμε και εμείς συνηθίσει αυτά τα φαινόμενα που αν τα γνώριζαν οι ψηφοφόροι τα απορούσαν και τα εξαρκιζόταν μαζί μας. Αν έρθουμε στην ουσία, πριν τρία χρόνια υιοθετήσαμε την έκθεση μου για το οικιακό προσωπικό και προσωπικό φροντίδας. Και παρά ότι το τονίστηκε με κάθε τρόπο και προς όλες τις πλευρές ότι ο κλάδος χρειάζεται ρύθμιση και προστασία, Δυστυχώς δεν έχουμε δει την αντίστοιχη νομοθετική πρόταση ακόμα. Το γεγονό ότι σήμερα συζητάμε ένα ψήφισμα και όχι μια πρόταση οδηγία ή κανονισμού δείχνει ότι περιοριζόμαστε σε ευχές και δεν προχωρούμε σε δεσμευτικές πολιτικές στο θέμα των υπηρεσιών φροντίδας και μιλάμε για τον σκληρό πύρινα του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους, για την φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικία των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία, το βάρος της φροντίδας πέφτει στις πλάτες των γυναικών και τις εμποδίζει να έχουν ίση πρόσβαση στην εργασιακή και κοινωνική ζωή. Ξεκινάμε την δουλειά μας στην έκθεση αυτή καλούμενοι να διαχειριστούμε μια παταγώδη αποτυχία. Στο προσχέδιο της έκθεση που συζητάμε αναφέρεται ότι οι στόχοι που έχουν οριστεί από το 2002 στη Βαρκελόνη για την βρεφονιπιακή και προσχολική μέρημνα των παιδιών κάτω των 6 ετών, οι στόχοι έχουν επιτευχθεί μόνο σε 12 από τα 28 κράτη-μέλη. Και μόνο αυτή η αποτυχία θα αρκούσε για να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να καλύψουμε το πρόβλημα με ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα. Και σε τι οφείλεται αυτή η μεγάλη αποτυχία που έχει επιβιώσει τη θέση των γυναικών την τελευταία δεκαετία. Νομίζω ότι η έκθεση πρέπει να λέει τα πράγματα με το όνομά της. Την τελευταία δεκαετία έχει γίνει αληθινή σφαγή στις κοινωνικές δαπάνες όλων των κρατών μελών με τις ευλογίες της Κομισιόν και του Συμβούλιο στο όνομα της κρίσης και των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Αυτό που λέμε λιτότητα δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο δεν είναι μια ιδεολογική αιμονή της αριστεράς, όπως μπορεί να σκέφτονται κάποιες άλλες πολιτικές ομάδες. Είναι συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις που πάρθηκαν τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στις χώρες που πέρασαν από μνημόνια όπως η Ελλάδα και μεταφράζονται σε λιγότερες βρεφο νηπιακούς σταθμούς, λιγότερες δομές φροντίδας, ηλικιωμένους και αρρώστους, λιγότερες κριτικές δαπάνες που θα βοηθήσουν τις εργαζόμενες γυναίκες να μοιραστούν το βάρος της φροντίδας με καταρτισμένους βοηθούς ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες εργασίας. Είναι τεράστια οπισθοδρόμηση για την Ευρώπη και για την κατάσταση των γυναικών, το γεγονό ότι γίνονται το υποκατάστατο του κοινωνικού κράτους που ακροτηριάζεται σχεδόν σε όλες τις χώρες. Και αυτό η έκθεση μας πρέπει να το λέει ανοιχτά. Φυσικά και πρέπει να βρούμε τρόπους να αναγνωρίσουμε την ανεπίσημη φροντίδα σε παιδιά ηλικιωμένους και άτομα αναπηρία και να υποστηρίξουμε τους άτυπους φροντιστές, ιδιαίτερα τις γυναίκες. Αλλά η προτεραιότητα μας πρέπει να είναι να, να αποκαταστήσουμε το πετσοκόμενο κοινωνικό κράτος. Σε αυτό το σημείο θέλω να υπογραμμίσω μια βασική διαφωνία με το σχέδιο έκθεσης. Σε αρκετά σημεία τη τονίζει ότι η πρόσβαση σε ποιοτικέ υπηρεσίε φροντίδα είναι κυρίω θέμα ατομική επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικά είδη φροντίδα, δημόσια ή ιδιωτική. Είναι τεράστιο λάθο. Η βασική μα κατεύθυνση πρέπει να είναι η δημιουργία και η ενίσχυση ενό αξιόπιστου δικτύου δημόσιων και κοινοτικών υπηρεσιών φροντίδα, και όχι η δημιουργία μια κερδοσκοπική αγοράς φροντίδας. Αυτή η αγορά έχει δοκιμαστεί ήδη ιδιαίτερα στη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων και έχει λειτουργήσει ως παράγοντας αποκλεισμών και ανισοτήτων εις βάρος των φτωχότερων οικογένειων και γενικών. Ο ιδιωτικό τομέα φροντίδα πρέπει να λειτουργήσει μόνο επικουρικά και υπό αυστηρή υποπτία και όχι ανταγωνιστικά προς το δημόσιο τομέα. Θέλω να δηλώσω την υποστήριξή μου στη θέση της εισηγήτρια να περιληφθούν στην διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξάμεινου η παρακολούθηση δεδομένων για την φροντίδα ηλικιωμένων και αναπήρων για την ακρίβεια πρέπει να υποστηρίξουμε την ένταση και αυτών των στοιχείων σε ένα σύνολο από κοινωνικούς δείκτες. Από την ανεργία μέχρι την ισότητα των γυναικών και από την ποινική φτώχεια μέχρι την κατάσταση της δημόσιας υγείας. Και σε αυτό πρέπει να συντονιστούμε καλά με άλλες εκθέσεις που συζητούνται αυτή την περίοδο στη δική μας και σε άλλες επιτροπές. Τελειώνοντας, επισημαίνω ότι η έκθεση μας δίνει την ευκαιρία να καλύψουμε κενά και αντιφάσεις της νομοθεσίας μας. Ένα μόνο παράδειγμα. Στο σχέδιο έκθεση η συγκήτρια επιθυμίζει την ανάγκη να τεθούν ως στόχοι η προοδευτική παράταση της γονικής άδειας, η προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων της γυναίκας φροντίστριας και η έναντι της απόλυσης. Σας θυμίσω την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δημιούργησε μια τεράστια νομική θρύπα. Οι έγκυες γυναίκες δεν προστατεύονται στις σωματικές απολύσεις. Είναι μια τεράστια οπισθοδρόμηση είναι μια τεράστια οπισθοδρόμηση. Και ως Ευρωβουλευτές, ιδιαίτερα ως Επιτροπή Γυναικών, πρέπει να έχουμε την φιλοδοξία να κλείσουμε αυτή τη τρύπα το τοχύτερο δυνατό. Σας ευχαριστώ. Θα επανέλθω με τις τροπολογίες που θα καταθέσω στο σχέδιο έκτασης. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κούνεβα και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το σχέδιο έκθεσης, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και που αναφέρει κάποια από τα θέματα πάνω στα οποία εργαζόμαστε πολύ εντατικά και εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, από πέρσι τον Απρίλιο που υιοθετήσαμε την οδηγία για την εξισορρόπηση ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου. Αρκετές από τις προτάσεις της έκθεσης ε, είναι πρωτοβουλίες, είναι μέτρα τα οποία αναφέρουμε στην ανακοίνωσή μας. Συμμεριζόμαστε μαζί σας ε, λοιπόν την άποψη ότι είναι σημαντικό να εξετάσουμε την διαθεσιμότητα ε, και την πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας για να μπορέσουν να συνδυάσουν τον επαγγελματικό και τον ιδιωτικό βίο. Νομίζω επίσης ότι είναι σημαντικό να γίνει η σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτό ήταν πιο σαφές και κατά το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Λαμβάνουμε υπόψη μας όμως τις προτάσεις που έχετε υποβάλει για περαιτέρω ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ επίσης για την σύνδεση που γίνεται με την πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου για οι υπηρεσίες οικονομικά προσβάσιμες ε, για την ε, πρώτη παιδική ηλικία και την ε, εκπαίδευση. Διαθεσιμότητα, οικονομική προσβασιμότητα και υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών. Καθώς και οι συνθήκες εργασίας των φροντιστών είναι θέματα πολύ σημαντικά. Ε, περιμένουμε λοιπόν ε, να δούμε την περαιτέρω εξέλιξη των προτάσεων. Επίσης, επικροτούμε ε, το, την ιδιαίτερη εστίαση σε παιδιά από μειονεκτικές οικογένειες. Για τα παιδιά αυτά είναι πολύ σημαντική η φροντίδα. Εκτιμούμε επίσης την προοπτική που παρακολουθεί το σύνολο της ε, ζωής, ε, δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στα παιδιά. Ε, πάντως, περιμένουμε με αγωνία να δούμε τα επόμενα βήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στην κυρία Πιετικάινεν πάλι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και οδησυσυγητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις τους. Προσλέπω στη συνεργασία πάνω στο θέμα αυτό. Περιμένω λοιπόν τις τροπολογίες σας και άλλες παρατηρήσεις για να έχουμε μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ανακοινώσω την ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 10 ε, Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. 12 Ιουλίου, 6 το απόγευμα. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, ε, το σημείο 10. Προεδρία του Συμβουλίου. Παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρίας του Συμβουλίου από τη Ιουλιάνε Μπόκνερ Στράους, Ομοσπονδιακή Υπουργό στην Ομοσπονδιακή Καγκελαρία Γυναικών, Οικογένειας και Νεολαίας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συντονιστές, Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, ε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση να σας παρουσιάσω σήμερα στην Επιτροπή Γυναικών της προτεραιότητες ε, της Αυστριακής Προεδρίας. Πιστεύω ότι όλοι συνειδητοποιούμε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ένα περιβάλλον με διάφορες προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Από τη μία πλευρά ελπίζουμε σε ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ε, για το Brexit, αλλά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών μας δείχνουν ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορες προκλήσεις. Από την άλλη πλευρά, Πρέπει να διαπραγματευτούμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κάτι που επίσης αποτελεί πρόκληση. Ε, επίσης, λίγη η νομοθετική θητεία και υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα τα οποία θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Το δικό μας σύνθημα είναι Ευρώπη που προστατεύει τα τελευταία χρόνια. Είδαμε διάφορες κρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να μεταφέρουμε και πάλι το μήνυμα στους πολίτες μας ότι η Ευρώπη είναι ασφαλής τόπος και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να λύνει προβλήματα προς συμφέρον των πολιτών μας. Θέλουμε ασφάλεια και ειρήνη και αυτό θα πρέπει να δώσουμε στην Ευρώπη. Θέλουμε να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σημαντικά θέματα και γι' αυτό επαναλαμβάνω το σύνθημα της Αυστριακής Προεδρίας «Η Ευρώπη που προστατεύει». Τρεις προτεραιότητες έχουμε θέσει ασφάλεια και καταπολέμηση της παράνομης ε, μετανάστευσης, αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων, διασφάλιση της ευημερία και της ανταγωνιστικότητας με την ψηφιοποίηση και σταθερότητα στις γειτονικές χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης. Επίσης, θέλουμε να ενισχύσουμε την αρχή της επικουρικότητας. Χρειαζόμαστε ενίσχυση της εμπιστοσύνης και πρέπει να βρισκόμαστε κοντά στο πολίτη. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί στα βασικά ερωτήματα, ενώ τα ε, λιγότερο σημαντικά θα πρέπει να ε, αντιμετωπιστούν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Θέλουμε λοιπόν ε, λιγότερα αλλά πιο αποτελεσματικά. Πρόοδος είναι δυνατό να σημειωθεί μόνο εάν τα κράτη-μέλη ε, ενεργήσουν ενωμένα. Η Ευρώπη θα προσπαθήσει να οικοδομήσει γέφυρες. Θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε την ενότητα της Ευρώπης. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στους στόχους και τις πρωτοβουλίες μας όσον αφορά τις γυναίκες. Η ισότητα των δύο φύλων είναι σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το είδαμε στο Ευρωβαρόμετρο του 2017, το 91% ε, των πολιτών απάντησαν ότι θεωρούν ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι πολύ σημαντικό στοιχείο ε, για μια δίκαιη και ευμερούσα ε, κοινωνία. Ενώ το 84% είπαν ότι η δικαιοσύνη είναι σημαντική για αυτούς τους ίδιους ε, όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων. Ε, η ισότητα των δύο φύλων θεσπίζεται και στη συνθήκη. Αναφέρεται ως ρητό καθήκον και αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γυναίκες και οι άντρες θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες. κάτι που ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για όλα τα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει κοινή στρατηγική για ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων. Υπήρχε μια τέτοια στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τώρα πια όμως δεν υπάρχει και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε στο μέλλον, να δώσουμε περισσότερη προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Η ισότητα ανδρών και γυναικών θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως άλλωστε βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις και από την ε, μελέτη, πολλοί πολίτες θεωρούν ότι θα πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα και να υπάρχει πολιτική στρατηγική. Μαζί με την Εστονία και τη Βουλγαρία, ε, τους εταίρους μας στο τρίο των Προεδριών, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό και έχουμε υπογράψει κοινή δήλωση για την ισότητα των δύο φύλων. Οι, κοινωνικές, οι οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις ε, έχουν αυξηθεί και σε πολλά κράτη-μέλη όπως και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρείται συχνά ότι ε, έχουμε πετύχει τα πάντα στον τομέα της ισότητας, αλλά απέχουμε πολύ από κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τον διάλογο για την ισότητα των ε, δύο φύλων μία διάσκεψη έχουμε οργανώσει ε, και θέλουμε να θέσουμε τα ερωτήματα ε, τι μορφή θα πρέπει να έχει η ισότητα στο μέλλον, τι ιδέες και ανάγκες έχουν ιδιαίτερα οι νέοι στην Ευρώπη, τι μέτρα είναι απαραίτητα για να πετύχουμε τον στόχο αυτό της ισότητας ε, των άνδρων και γυναικών. Μετά έχουμε τη διάσκεψη ε, ισότητα των δύο φύλων και νεολαία που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και χαίρομαι πολύ που ήδη κάποιοι από εσά έχετε δηλώσει συμμετοχή και θα παρευρεθείτε στην διάσκεψη αυτή για να συζητήσουμε μαζί τα θέματα. Ασχολούμαστε λοιπόν με το θέμα αυτό και θα υπάρξει διαδραστική ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε νέους ε, υπουργούς, ε, υψηλόβαθμους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπειρογνώμονες από μη κυβερνητικές οργανώσεις και ε, ανθρώπους από τις διοικήσεις των κρατών μελών. Θα έχουμε λοιπόν ομαδική συζήτηση για δια τομεακή αλλά και για διαγενειακή συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσά ήδη έχετε δηλώσει συμμετοχή. Ε, όσο περισσότεροι βρεθούμε στη Βιέννη για τη διάσκεψη αυτή, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία μπορούμε να περιμένουμε να έχει. Είναι σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή σας για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των δύο φύλων να ε, εκπροσωπείται στην διάσκεψη αυτή για να μπορέσουμε να κινήσουμε τα πράγματα στην Ευρώπη και να θέσουμε και πάλι την ισότητα των δύο φύλων ως προτεραιότητα. Για μένα, ως Υπουργό Νεολαίας, είναι πολύ σημαντικό το θέμα και των νέων ανθρώπων. Ε, μαζί με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεότητας και τον ε, αντίστοιχο ε, Αυστριακό Οργανισμό, Θέλουμε να ακουστεί η φωνή των νέων, θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή τους και όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων. Θα πραγματοποιηθούν προπαρασκευαστικά εργαστήρια σε σχολεία, στο Στρασβούργο, στις Βρυξέλλες και σε διάφορες πόλεις στην ε, Αυστρία. Έτσι ακούμε ποιες είναι οι ανάγκες των νέων ανθρώπων όσον αφορά την ισότητα ανδρών και γυναικών. Οι απόψεις ε, είναι τολμηρές και πολύμορφες και θέλουμε αυτό το όραμα να το θέσουμε στο επίκεντρο της διάσκεψης για την ισότητα των δύο φύλων. Άλλο σημαντικό θέμα για μας είναι οι ευκαιρίες που παρέχει η ψηφιοποίηση στα αγόρια και στα κορίτσια. Στο επίκεντρο του διαλόγου για την ισότητα βρίσκεται το θέμα της ψηφιοποίησης, σε κάτι που έχει απασχολήσει και το τρίο ε, της Προεδρίας, δηλαδή την Αυστρία μαζί με την ε, Εστονία και την Βουλγαρία. Με το κλείσιμο λοιπόν αυτού του τρίου της Προεδρίας και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για την Ισότητα θέλουμε να εξετάσουμε τις ευκαιρίες και τους κινδύνους της ψηφιοποίησης για τα κορίτσια και τα γόρια. Θέλουμε έτσι να εξετάσουμε τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται και μέσω της πολιτικής συμμετοχής μέσω των ψηφιακών μέσων και θέλουμε να εξετάσουμε εάν τα γόρια και τα κορίτσια υποφελούνται εξίσου από τις ευκαιρίες που παρέχει η ψηφιοποίηση. Επίσης, όσον αφορά την επιγραμμική βία, θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό που είναι η σκοτεινή πλευρά της ψηφιοποίησης. Θέλουμε όλα αυτά να αποτελέσουν βάση για συμπεράσματα όσον αφορά την ψηφιοποίηση και την νεολαία τα τελικά συμπεράσματα ε, θα συμπεριλαμβάνουν και αναθεώρηση της δήλωσης του Πεκίνου και της σχετικής πλατφόρμας δράσης. Θέλουμε να δώσουμε μια θετική κατεύθυνση στη συζήτηση. Πώς μπορούμε λοιπόν να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια για να ε, ε, εκμεταλλευτούν ε, τα, τις ευκαιρίες που παρέχει η ψηφιοποίηση. Πώς μπορεί η ψηφιοποίηση να προσανατολιστεί ώστε να ενισχύσει τις ευκαιρίες ε, αγοριών και κοριτσιών και επίσης να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ε, με θετικό τρόπο τους κινδύνους της ψηφιοποίησης. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε προτάσεις πάνω στα θέματα αυτά gender mainstreaming, ενσωμάτωση της διάστασης ε, της ισότητας ε, των δύο φύλων. Και αυτό είναι θέμα που απασχολεί την αυστριακή κοινωνία και επίσης έχει συμπεριληφθεί ως προτεραιότητα στο 18μηνο του τρίου των Προεδριών. Και κατά την διοργάνωση έχει ληφθεί υπόψη το θέμα αυτό και κατά την προετοιμασία της Αυστριακής Προεδρίας είχαμε στην Αυστρία διπουργική ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Τα Υπουργεία, το Κοινοβούλιο, το στατιστικό, η Στατιστική Υπηρεσία και τα κρατήδια μας έχουν υποβάλει απόψεις, έχουν ανταλλάξει απόψεις σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης των δύο φύλων μαζί με την ε, Γραμματεία του Συμβουλίου. Έχουμε εξετάσει ε, δείγματα βέλτιστων πρακτικών. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό οι συγκεκριμένοι ε, στόχοι να συνδέονται με συγκεκριμένα μέτρα. Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τις εμπειρίες που έχουμε στον τομέα αυτών ε, καθώς και τις εμπειρίες που θα ε, συγκεντρώσουμε κατά τη διάρκεια του επόμενου εξαμήνου και ε, να τις μεταφέρουμε στο επόμενο τρίο προεδριών για να συνεχιστούν οι προσπάθειες. Έχουμε σχέδιο οδηγίας για την εξισορρόπηση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Το θέμα αυτό αποτελεί σημαντικό τμήμα της κοινωνικής και πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης και είναι και σημαντικό θέμα για ε, το κάθε άτομο. Θα πρέπει λοιπόν να διευκολυνθεί ο συνδυασμός ε, οικογενειακής και επαγγελματική ζωής, λαμβάνοντας υπόψη και τη δημογραφική αλλαγή και τις αλλαγές στην αγορά εργασία. Χαίρομαι λοιπόν που μπορώ να σας ενημερώσω ότι στις 21 Ιουνίου το Συμβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση ξεκινάμε διαπραγματεύσεις. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο, μόλις καταλήξετε κι εσείς σε πρόταση και προσλέπω στην, ε, στον καλό διάλογο και την επικοδομητική συνεργασία με το Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε σε ισορροπημένη λύση. Τα κράτη-μέλη συμφωνούν μεταξύ τους ότι μέτρα για βελτίωση ε, του συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα πρέπει όμως να φροντίσουμε να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικές ιδιαιτερότητες, ώστε τα μέτρα να μπορέσουν πράγματι να εφαρμοστούν σε όλα τα κράτη-μέλη. Προσχώρηση στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για μένα ως Αυστριακή το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Αυστρία ήταν ένα από τα πρώτα κράτη που εφήρμοσαν τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και είμαστε και έχουμε ήδη εξετάσει και τον ε, αντίκτυπο. Η καταπολέμηση κάθε μορφής βίας εις βάρος γυναικών και κοριτσιών ε, είναι ένα σημαντικό θέμα που συνδέεται και με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε λοιπόν κάθε είδος βίας ε, εις βάρος ε, των γυναικών. Η βία δεν έχει χώρο στην Ένωση. Θα ήθελα επίσης να πω ότι και τα 28 κράτη-μέλη ήδη έχουν υπογράψει τη σύμβαση, τα 18 εκ των οποίων την έχουν επικυρώσει. Τον ε, Μάιο του 2017 ξεκίνησε η διαδικασία. Η Προεδρία μας ε, θα ασχοληθεί με την ολοκλήρωση του θέματος αυτού και θέλουμε να εκπονήσουμε κώδικα δεοντολογίας για την εφαρμογή της σύμβασης. Θα ήθελα να αναφερθώ στο σχέδιο οδηγίας για τις γυναίκες σε ηγετικές ε, θέσεις. Σε στα διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων. Έχει μπλοκάρει το θέμα και γι' αυτό πέρσι στο Συμβούλιο δεν είχαμε ε, σχετικές συζητήσεις. Η Αυστρία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση ε, και θα λάβει υπόψη και την ε, στάση των άλλων κρατών μελών. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην οδηγία κατά των διακρίσεων. Οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο είναι δύσκολες, διότι απαιτείται ομοφωνία στο θέμα αυτό. Και δεν υπάρχει συμφωνία ούτε όσον αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων. Από το 2008 και μετά εξετάζεται το θέμα. Ε, υπό την δική μας Προεδρία θα συνεχιστούν οι σχετικές συζητήσεις στην ομάδα εργασίας. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε θερμά κύριε Υπουργέ για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων τη Αυστριακή Προεδρία. Παίρναμε στη συζήτηση. Η κυρία Κοζουόφσκα. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Υπουργέ, κύριε και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την εκπρόσωπο της Προεδρία Προεδρίας ε, για την παρουσίαση και τι δηλώσει τη για την στην εκτίμηση τη διάσταση του φίλου στι ευρωπαϊκέ πολιτικέ και για τη συνθήκη τη Κωνσταντινούπολη. Ήθελα να πω ότι συμφωνώ μαζί σα, κύριε Υπουργέ, ότι είναι πολλά τα επιτεύγματά μα ε, ω προ την ισότητα των φίλων, Ναι, μεν, αλλά τα επιτεύγματα αυτά βρίσκονται σε επίπεδο διακηρυκτικό. Ε, τα περισσότερα είναι πολιτικέ διακηρύξει. Αν δεν περάσουμε από τις διακηρύξεις στις νομοθετικές προτάσεις, ε, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτή η νομοθετική ε, μεταγραφή των διακηρύξεων ε, μας ενδιαφέρει. Οπότε και το νομοθετικό σκέλος ε, μας ενδιαφέρει, αλλά πρώτα απ' όλα η εφαρμογή της εγκριθής νομοθεσίας. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο. Άλλο θέμα, το πακέτο για τον συνδυασμό ιδιωτικού και επαγγελματικού βίου. Ποια είναι η θέση της Αυστριακής Προεδρίας για τα ζητήματα αυτά. Φυσικά εκτιμώ και σέβομαι τη θέση του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου, αλλά δεν κρύβω την απογοήτευσή μου για την υπερβολικά μετριοπαθή κοινή θέση του Συμβουλίου, ε, πολύ λιγότερο φιλόδοξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ε, άδεια πατρότητας ε, την εννιά ημέρη. Ε, δυστυχώς δεν ε, ενέκρινε κανένα άλλο τμήμα της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Συμβούλιο και άφησε όλα τα ζητήματα στην εθνική διακριτική ευχέρεια. Οπότε τα πράγματα θα μείνουν ως έχουν στις περισσότερες χώρες που οι άδειε πατρότες και μητρότες είναι συνήθως άνευ αποδοχών στα περισσότερα κράτη-μέλη. Ε, επίσης, άλλο θέμα είναι η μεταβιβασιμότητα της ε, άδειας, ε, της γονικής άδειας. Αν όμως γίνει μεταβιβάσιμη άδεια και μπορεί η άδεια πατρότητας να μεταφέρεται στη γυναίκα ως άδεια μητρότητας, τότε θα την αξιοποιούν περισσότερο την άδεια οι γυναίκες, οπότε η υποεκπροσώπησή τους και η απουσία τους από την αγορά εργασίας θα διονυστεί. Ελπίζω στη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας ε, να μεταπιστεί κάπως το Συμβούλιο, να αλλάξει θέση και να ε, φανεί πιο διαλλακτικό στις συζητήσεις. Γιατί δυστυχώς ε, οι δικές μας προτάσεις απέχουν παρασάγκας από τις προτάσεις του Συμβουλίου. Θα πρέπει να ε, προτείνεται μεγαλύτερη σύγκληση έγινε. Χαίρομαι επίσης για, το προ... τις προτάσεις ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση και την πρόσβαση των νέων σε θέματα ε, ψηφιοποίησης κυρίως των κοριτσιών. Γιατί θα πρέπει να προσελκύσουμε τις γυναίκες, τα κορίτσια και τις γυναίκες ε, στους νέους τομείς και τις ψηφιοποίησεις ώστε να μπορέσουν και αυτές να εντοχθούν στα νέα προγράμματα βιομηχανοποίησης 4.0. Επίσης, ε, θέλουμε προγράμματα που θα στοχεύουν ιδιαίτερα στα έφηβα κορίτσια, γιατί από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό. Και τέλο, για τη διάσκεψη που θα πραγματοποιήσει η Αυστρία ε, για την ισότητα. Ελπίζω να έχουμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε και τι λεπτομέρειε τη σχετική διάσκεψη. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, κυρία Κοζόφσκα. κυρία Μλίναρ. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ για την παρουσίασή σας και που βρήκατε το χρόνο να έρθετε εδώ να συζητήσετε μαζί μας. Χθες βρισκόμουν στην Επιτροπή Εσωτερικών όπου οι Επιτροπές Κίκλ και Μόζερ ε, παρουσίασαν το πρόγραμμα της Ευρώπης που προστατεύει και είπα και το επαναλαμβάνω σήμερα ότι η Ευρώπη που προστατεύει θα πρέπει να βασίζεται ε, στι αξίες της Ευρώπης. Και ήθελα να το τονίσω αυτό διότι πότε πότε ξεχνιέται. Ε, συζητάμε εντό ενό πλαισίου ασφαλεία, αλλά δεν ξέρουμε τι κατεύθυνση θα πάρει τελικά. Σας ευχαριστώ που τονίσατε το θέμα της ενσωμάτωσης της διάστασης ε, των ε, δύο φύλων. Είμαι η συγγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό και είμαι στη διάθεσή σας για συζήτηση και συνεργασία στο θέμα αυτό. Όσον αφορά την ε, Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, επικροτώ τη θέση σας πάνω στο θέμα αυτό. Ποια είναι η θέση της Αυστριακής Προεδρίας Όσον αφορά τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, πώς μπορείτε να τα κινητοποιήσετε ώστε τελικά να έχουμε επικύρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που είναι απαραίτητο. Και τέλος, μια δύσκολη ερώτηση. Ε, αν γίνει αναπροσαρμογή της οικογενειακής ενίσχυσης στην Αυστρία, Αυτό θα επηρεάσει τις ε, γυναίκες από άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Έτσι θα γίνει διάκριση εις βάρος των γυναικών αυτών. Γνωρίζουμε ότι η πρόταση αυτή ε, θα αντίκειται στο ευρωπαϊκό δίκαιο ε, και η σχετική απόφαση του Κοινοβουλίου της Αυστρίας έχει καθυστερήσει, διότι φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Εσείς εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι βήματα θα κάνετε για να καταλήξετε σε μια συνολική ευρωπαϊκή θέση. Εάν η Αυστριακή Προεδρία ε, υιοθετήσει πράξη που θα οδηγήσει σε σε διαδικασία παράβασης της συνθήκης. Ε, πώς το βλέπετε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κυρία Υπουργέ στην Επιτροπή για τα δικαιώματα των γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας. Θα ξεκινήσω από κάτι θετικό. Ήταν θετική έκπληξη το πόσο αναλυτικά μας παρουσιάσατε το περιεχόμενο του προγράμματος. Διότι δεν σας κρύβω, ήμουν απογοητευμένη που το θέμα της πολιτικής γυναικών και της ισότητας ήταν ένα θέμα που αναφερόταν μόλις ε, ε, σύντομα στην σελίδα 42 του προγράμματος Αυστριακής Προεδρίας, ε, ενώ στο πρόγραμμα του Τρίο έπιανε πιο πολύ χώρο. Πάντως, σας ευχαριστώ πολύ που μας παρουσιάσατε τόσο αναλυτικά το πρόγραμμα της Προεδρίας σας στον τομέα αυτό. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε αυτό που είπε η προλαλή σας Αγγέλικα Μίνα. Ευρώπη που προστατεύει. Όταν ε, διαβάζουμε στον τύπο ε, αυτά που γράφονται για την Αυστριακή Προεδρία, βλέπουμε μόνο ε, το θέμα της ε, μετανάστευσης και ε, της προστασίας των εξωτερικών συνόρων. Ενώ υποεκπροσωπούνται, εάν εμφανίζονται καν τα θέματα ισότητας των, των γυναικών. Κατά το εξάμεινο της Αυστριακής Προεδρίας, θα έχουμε την τελευταία ευκαιρία πριν τις ευρωεκλογές για να θέσουμε την κατεύθυνση για μια Ευρώπη δικαιωμάτων των γυναικών. Είναι λοιπόν μεγάλη η ευθύνη της Αυστριακής Προεδρίας. Όπως και οι προλαλήσασες, ε, θα ήθελα να αναφερθώ στην κοινωνική Ευρώπη και την σημασία της απασχόλησης διότι περιμένουμε πολλά από την Αυστριακή Προεδρία. Ερώτηση καταρχάς για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βρίσκω κρίμα που ο Υπουργός ε, κύριος Λούγκερ δεν θα εμφανιστεί αυτή την εβδομάδα στην Επιτροπή Προϋπολογισμού για να αναφερθεί στο θέμα του προϋπολογισμού, διότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικά θέματα της Προεδρίας και έχει μεγάλη σημασία και για τις γυναίκες και για την κοινωνική Ευρώπη. Στην Επιτροπή Γυναικών την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια ακρόαση για τον προϋπολογισμό και τη διάσταση του φύλου στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και καταλήξαμε στο στρομακτικό συμπέρασμα ότι δεν αναφέρεται καν το θέμα αυτό, δηλαδή έχουμε οπισθοδρόμηση σε σχέση με το ισχύον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ρωτώ λοιπόν, εσείς ως, γραμματεία, ως Προεδρία του Συμβουλίου, τι θα κάνετε για να συμπεριλαμβάνετε το θέμα της διάστασης των φύλων στον προϋπολογισμό. Και επίσης, ε, γιατί να μην, είναι, γιατί να μην συνεχίσει να είναι οριζόντιο θέμα στα διαρθρωτικά ταμεία. Επίσης, το θέμα της βίας κατά των γυναικών αναφέρθηκε ήδη η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Πώς μπορεί να πρικοδοτηθεί καλύτερα ένα πρόγραμμα όπως το Δάφνη και να υπάρξει ξεχωριστή γραμμή του προϋπολογισμού. Και επίσης, όπως η προλαλή βρίσκω και εγώ ανησυχητικό ότι η Αυστρία ε, επικρίνει το ευρωπαϊκό δίκαιο και μάλιστα με τρόπο που απειλεί τις γυναίκες όπως είναι η αναπροσαρμογή των οικογενειακών επιδομάτων αλλά και πώς βλέπετε το 12ωρο που θα εισαχθεί στην Αυστρία. Πώς ε, βλέπετε αυτά να συνάδουν με ε, τα δικαιώματα των γυναικών και το ισχύον δίκαιο. Ευχαριστώ Κύριε Στοσίνσκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ε, ασθενίζομαι πολλά θέματα, όπω η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και κυρίως ε, των ε, νερών κοριτσιών. Και χαίρομαι που η Αυστρία έχει ειδικό υπουργό για την οικογένεια από τότε που ανέλαβε ο Μακρό, καταργήθηκε αυτό το Υπουργείο στην Γαλλία. Κρίμα για μας. Μπράβο σε εσά. Τώρα, σήμερα το πρωί είχαμε στην Επιτροπή Γυναικών μία συζήτηση μετά από παρουσίαση που μας έκανε ε, η οργάνωση ε, Open Society, Ανοιχτή Κοινωνία, του δισεκατομμυριούχου γκρου George Σόρος θέμα ήταν το, τα Ισλαμικά, ε, Ισλαμικοί δημα, δηματολογικοί κώδικες, ε, όπως το η Μαντήλα. Η μαζική μετανάστευση που έχουμε δεχτεί στην Ευρώπη δημιουργεί ένα όλο και πιο επικίνδυνο πρόβλημα διαχωρισμού των επιμέρους κοινοτήτων, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Και έχουμε όλο και μεγαλύτερη παρουσία ε, δημ μουσουλμανικών ενδυμάτων, κυρίως γυναικείων. Στη Γαλλία απαγορεύονται αυτά στους δημόσιους χώρους, αλλά παρόλα αυτά πολλοί μουσουλμάνοι χρησιμοποιούν αυτόν τον περιορισμό για να προωθήσουν ε, τις ε, διεκδικήσεις τους. Ποια είναι η άποψη της Αυστρίας ε, για το θέμα αυτό, το, της μαντήλας και των μουσουλμανικών η κυρία Ρωσινιόλα, επί Αλάν, μιλούσαν για κίνδυνο εγκλωβισμού του σώματος των γυναικών σε ένα ένδυμα και κυρίως ε, η χρησιμοποίηση αυτού του Ισλαμικού ακτιβισμού υπέρ της ιδέας του πολιτικού Ισλάμ. Σας ευχαριστώ κυρία Μορβάη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ και σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή μας και μας παρουσιάσατε τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας. Μου άρεσε ιδιαίτερα η προτεραιότητά σας ε, να ενισχύσετε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταπολεμήσετε την λάθρο μετανάστευση, την παράτυπη μετανάστευση. Ας μην γελιόμαστε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η προτεραιότητα αυτή έχει και μία διάσταση έμφυλη. Η προτεραιότητα αυτή της προστασίας, της ενίσχυσης προστασίας εξωτερικών συνόρων έχει ιδιαίτερη σημασία για τις γυναίκες της Ευρώπης. Και γιατί το λέω. Το λέω με βάση την εμπειρία μου. Παρόλο που είμαι Ουγγαρέζα και πολλοί λένε ότι στην Ουγγαρία εσείς δεν έχετε καμία πείρα με τη μετανάστευση. Όχι, σας διαβεβαιώνω ότι έχουμε και εμείς εμπειρία με τη μετανάστευση. Στις αρχές του 2015, εγώ ε, που είμαι δικηγόρος ειδικευμένη στα δικαιώματα των γυναικών και ευρωβουλευτής, προσεκλήθη σε ε, στα σύνορα της Ουγγαρίας που είχαμε μαζική άφηξη μουσουλμάνων μεταναστών. Κάτι που άλλαξε ριζικά τη ζωή των ε, γυναικών σε εκείνη την αγροτική κοινότητα. Υπήρχε φόβος ε, για παραβίαση της αξιοπρέπειάς τους και η καθημερινότητα των τόπιων γυναικών άλλαξε ριζικά και μάλιστα προς το χειρότερο σε αυτή την ε, περιφέρεια. Μην μας λέτε λοιπόν ότι δεν έχουμε πείρα με την μετανάστευση. Οι περισσότεροι πολιτικοί ζουν μια προνομιακή ζωή. Και φαίνεται α, ε, κοφεύουν στα αιτήματα των γυναικών που υφίστανται τα δυνά της μετανάστευσης. Και ποια είναι αυτά τα αποτελέσματα. Ε, οι άνδρες αυτοί, οι μετανάστες, ε, έχουν γεννηθεί σε πολύ διαφορετική κουλτούρα και γεννήθηκαν και ανατράφηκαν πιστεύοντας ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετικό ρόλο από αυτό που πιστεύουμε εμείς ότι έχουν στην Ευρώπη. Και ε, μάλιστα αγχώνονται και εξοργίζονται όταν φτάνουν στην Ευρώπη αυτοί οι άνδρες και βλέπουν τις γυναίκες ακάλυπτες, με την κεφαλή ακάλυπτη, τις γυναίκες να δουλεύουν, να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής ε, μεταφοράς χωρίς να συνοδεύονται και γίνονται επιθετικοί αυτοί οι άνδρες μετανάστες. Αυτό βιώνουν λοιπόν οι γυναίκες στην Ευρώπη. Δεν μπορούν να γυρίσουν σπίτι ασυνόδευτες από τη δουλειά τους. Πρέπει να αναδιαμορφώσουν τη ζωή τους, την καθημερινή ζωή τους. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, το ποδήλατο για να πάνε από, τη μία, από το ένα σημείο της πόλης στην άλλη γιατί ε, έχουν υποστεί επιθέσει από δυσαρεστημένου άνδρε, δυσαρεστημένου με τον τρόπο ζωή του. τι κάνει μια γυναίκα σκέφτονται μόνη τη ένα ποδήλατο και υπάρχουν γυναίκε που μερικές φορές ε, έκαναν βόλτε το απόγευμα με τα παιδιά του, αλλά τώρα πια δεν τολμάνε, φοβούνται, γιατί έχουν δεχτεί και ελεκτικέ επιθέσει. <coughs> και είναι πολύ λεπτό το ζήτημα πια. Μπορούμε να περιμένουμε από την Αυστριακή Προεδρία κάποια αντιμετώπιση θα πρέπει καταρχήν να γίνει μια ευρεία εμβέλειας έρευνα για τις εμπειρίες που έχουν οι γυναίκες στην Ευρώπη από αυτή τη μαζική μετανάστευση. Εγώ ως πανεπιστημιακός και ως δικηγόρος που ασχολούμαι με τα γυναικεία δικαιώματα θα ενθάρρυνα και θα παρότρινα την Αυστριακή Προεδρία να κάνει τέτοια ε, εκτεταμένη έρευνα και χαίρομαι για το σύνθημά σας «Μια Ευρώπη που προστατεύει». Ελπίζω αυτό το σύνθημα της Αυστριακής Προεδρίας ε, να γίνει όντως πραγματικότητα, ώστε η Ευρώπη πραγματικά να προστατεύει τις Ευρωπαίες γυναίκες και τα κορίτσια της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ και καλή σας τύχη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό για την παρουσίαση που έκανε των θεμάτων της Αυστριακής Προεδρίας όσον αφορά την ισότητα των φίλων. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία ε, για την επίτευξη πρόοδου και θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Ε, καταρχάς, κάτι που σχετίζεται με την ισορροπία ιδιωτικής ζωής ε, και εργασίας. Είναι μία από τις προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου που αφορά την κοινωνική Ευρώπη για την υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα της Ευρώπης. Η Επιτροπή Γυναικών υιοθέτησε μια πολύ φιλόδοξη έκθεση και ελπίζω ότι θα εγκριθεί από την Επιτροπή Απασχόλησης αυτή. Ε, κυρία Υπουργέ, οι θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου είναι σαφείς βασίζεται σε αρχές. Όλες οι άδειες που θα εγκριθούν θα πρέπει να είναι επαμοιβή. η γονική άδεια δεν θα πρέπει να, να μεταφέρεται. ποια είναι η κατάσταση όμως στο Συμβούλιο, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στα κράτη-μέλη, πώς θα επηρεάσετε τα κράτη-μέλη ούτω ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή λύση. Πώς θα επηρεάσετε τα κράτη-μέλη, πώς θα ασκήσετε κάποια πίεση ούτως ώστε να ληφθεί μια απόφαση για την ισορροπία ιδιωτική ζωής και εργασιακής ζωής. Άλλη ερώτηση. Αυτή σχετίζεται με τη βία. Ήδη μίλησαν κάποιοι συνάδελφοι αυτό. Δέκα κράτη-μέλη δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ακόμα. Πώς θα πείσετε αυτά τα κράτη-μέλη να κυρώσουν την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Πότε θα επιτευχθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τη σύμβαση αυτή, την κύρωση της συμβάσεω της Κωνσταντινούπολης από πλευράς τη Ευρωπαϊκή Ανώσεως. Όσον αφορά α, την σχετική οδηγία, ήλπιζα ότι η Προεδρία της ε, Αυστρίας θα δραστηριοποιηθεί ούτως ώστε να προωθηθεί η οδηγία. Μετά την Προεδρία του Λουξεμβούργου κανείς δεν την επεξεργάστηκε. Θα κάνετε κάποια βήματα προόδου. Όσον αφορά τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, διότι αυτό θα ήταν πραγματικά σημαντικό βήμα για την ισότητα των φύλων. Ευχαριστώ. Θα σας δώσω το λόγο τώρα κυρία Υπουργέ, αν έχετε την καλοσύνη να σχολιάσετε τις ερωτήσεις των μελών. Έχετε το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Εν μέρη θα ε, απαντήσω στο βαθμό που είναι δυνατόν. Ήδη κατά την εισαγωγή μου είπα ότι είναι πολύ σημαντικό για μας η ισότητα των δύο φύλων να αποτελέσει και πάλι προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι το τέλος του 2015 υπήρχε στρατηγική για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Από το 2016 έως το 2019 Ισχύει ένα έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το οποίο σημαίνει ότι οι στόχοι δεν επιδιώκονται με ε, τον ίδιο βαθμό όσο και πριν. Εμείς θέλουμε λοιπόν και πάλι να έχουμε στρατηγική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μαζί προσπάθεια για να το πετύχουμε αυτό η ισορροπία οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Αυτό είναι ένα θέμα που αναφέρθηκε από αρκετούς από εσά. Προσβλέπουμε σε επικοδομητική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα κράτη-μέλη συμφωνούν μεταξύ τους σχετικά με τα όσα πρέπει να γίνουν για να βελτιωθεί η ισορροπία ανάμεσα στον οικογενειακό και τον επαγγελματικό βίο. Σε πολλά κράτη-μέλη Υπάρχουν πολύ καλά συστήματα ή συστήματα με σωστή χρηματοδότηση για την υποστήριξη της, του συνδυασμού οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη τα συστήματα αυτά ήδη λειτουργούν. Στην οδηγία αυτή λοιπόν και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει πάντα να προσέξουμε τα μέτρα στα διάφορα κράτη-μέλη να εφαρμοστούν και στην πραγματικότητα. Ο συνδυασμός επαγγελματικού και ε, ιδιωτικού βίου είναι πολύ σημαντικό για μένα να αποτελεί προτεραιότητα για να μπορέσουμε να επιφέρουμε βελτιώσεις στα κράτη-μέλη. Επίσης αναφέρθηκε από πολλούς από εσά η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Οι δύο, όπως είπα, και τα 28 κράτη-μέλη έχουν υπογράψει τη σύμβαση, ενώ 18 από αυτά την έχουν επικυρώσει κιόλας. Ενώ το περιεχόμενο θα το μετατρέψουμε σε κώδικα δεοντολογίας για την εφαρμογή της σύμβασης. Η Αυστρία ήταν από τα πρώτα κράτη-μέλη που υπέγραψαν και επικύρωσαν τη σύμβαση. Ήδη λοιπόν έχουμε εκπονήσει σχετική έκθεση που δείχνει ότι η Αυστρία εργάζεται πολύ καλά πάνω στα θέματα αυτά, απομένουν όμως πράγματα να κάνουν να, ε, πράγματα να γίνουν. Θέλουμε λοιπόν και τα άλλα κράτη-μέλη μαζί με μας να εφαρμόσουν την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, διότι το θέμα της βίας εις βάρος των γυναικών είναι πολύ σημαντικό θέμα. Επίσης, η προσχώρηση της, Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση θα αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για δικαιοσύνη ανάμεσα στα δύο φύλλα. Άλλωστε, η θεσμική βία αποτελεί και τη βάση για την ατομική βία. Θα βελτιωθεί έτσι και η διεθνής θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Μάιο του 2017 υιοθέτησε το Συμβούλιο και το περιεχόμενο της Σύμβασης και η Προεδρία μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα. Όσον αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η Αυστρία έχει μακρά παράδοση όσον αφορά το gender budgeting, η ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων στον προϋπολογισμό. Αυτό αποτελεί ήδη από το 2009 βασική έννοια στην Αυστρία. Η Αυστρία καταβάλει προσπάθειες ώστε σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα να κατανέμονται τα χρήματα, τα κονδύλια με τρόπο δίκαιο και για τα δύο φύλλα. Στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό από το 2013 εφαρμόζεται η σχετική αρχή. Οι διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα συνεχιστούν και υπό την Αυστριακή Προεδρία. Εδώ θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να υποφεληθεί το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη φυσικά το θέμα της διάστασης των δύο φύλων. Όσον αφορά τις θέσεις γυναικών σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, η Αυστριακή Προεδρία θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα αυτό και θα λάβει υπόψη τις θέσεις και των άλλων κρατών μελών. Από αυστριακής πλευράς μπορώ να σας πω ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2018 η Αυστρία έχει εφαρμόσει νομοθεσία σχετικά με τις θέσεις γυναικών σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων. Άλλο θέμα είναι η ενδυμασία των γυναικών. Εδώ θα σας αναφέρω την προσωπική μου θέση. Είναι σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση κράτους θρησκείας. Οι ενδυματολογικές επιλογές των γυναικών ε, θα πρέπει να γίνονται σεβαστές. Οι γυναίκες θα πρέπει να επιλέγουν οι ίδιες τι θέλουν να φορέσουν. Κατόπιν έχουμε το σύνθημά μας, η Ευρώπη που προστατεύει. Αυτό θέλουμε να το δούμε σε διάφορα επίπεδα και όχι μόνο όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση. Όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση και το θέμα των γυναικών μεταναστών που αναφέρατε κι εσείς, έχει ως εξής. Ε, θέλουμε να εμποδίσουμε την παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν σε αυτό, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε και αυτούς που χρειάζονται βοήθεια. Και δεν θα πρέπει τελικά οι διακινήτέ να αποφασίζουν ποιο θα ε, φτάσει στην Ευρώπη, αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν. Σημαντικό για όλους μας είναι να αποφύγουμε τους πολλούς θανάτους που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο και να έχουμε δίκαιες αποφάσεις σχετικά με το ποιος επιτρέπεται να φτάσει στην Ευρώπη και ποιος όχι. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις Ευρώπης. Α, όσον αφορά το οικογενειακό επίδομα, αυτό είναι εθνική υπόθεση, κατά τη γνώμη μου. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη με τα οποία συνομιλούμε εντατικά πάνω στο θέμα αυτό. Υπάρχουν και κάποια κράτη-μέλη που θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να γίνεται αναπροσαρμογή του, του επιδόματος. Θα πρέπει να καλύπτεται μέρος του κόστους των οικογένειών το κόστος αυτό διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Γι' αυτό ζητάμε να εξεταστεί τι μορφή έχουν οι διάφορες πρακτικές στα διάφορα κράτη-μέλη όσον αφορά το οικογενειακό επίδομα. Θα ήθελα όμως να αναφέρω ότι το θέμα αυτό αποτελεί αντικείμενο εθνικής διαπραγμάτευσης. Στον κανονισμό 883 συμπεριλαμβάνεται το θέμα αυτό, αλλά αυτό δεν είναι αρμοδιότητα ε, της δικής σας Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Μία σύντομη ερώτηση <coughs> για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Θα ήθελα να σας πω κύριε Υπουργέ ότι για το θέμα αυτό Έχω για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, παρακαλώ, για τον τιμάριθμο. Ε, θα ήθελα να σας πω ότι μαζί με την κυρία Σοβιέσκα υποβάλαμε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ερώτηση ήταν, η απάντηση ήταν κατηγορηματική, ότι τέτοιου είδους δράσεις ε, είναι απαράδεκτες. Ε, πάντως ο εργαζόμενο καταβάλει εισφορέ και στα πλαίσια αυτών των εισφορών ε, λαμβάνει επίδομα. Φυσικά διαφορετικά υπολογίζουν τα κάθε κρατημένη το ύψος του επιδόματο, οπότε έγιναν φαντάζομαι συζητήσει για τα θέματα αυτά και έχει εθνηθεί κάποια στάση στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ich darf hier noch θα ήθελα να ότι η εισφορά για το οικογενειακό επίδομα δεν, δεν γίνεται από τους εργαζομένους, αλλά από τους εργοδότες. Άσχετα δηλαδή από το αν ο εργαζόμενος έχει παιδί ή όχι, ο εργοδότης πρέπει να συνεισφέρει σε αυτό το ταμείο. Τα επιχειρήματα είναι πολλά. Γνωρίζετε ότι και στην ε, Βρετανία προτάθηκε αναπροσαρμογή των οικογενειακών ε, επιδομάτων. Αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Και για μένα είναι θέμα δικαιοσύνης. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει κατόφλι συχνά χαμηλό, δηλαδή 300 ευρώ, από το οποίο δεν πληρώνεται πια οικογενειακό επίδομα. Αυτό που ζήτησα λοιπόν είναι να εξεταστεί το θέμα αναλυτικά, ώστε να έχουμε δίκαιη μεταχείριση ώστε να μην ε, πρέπει να πληρώνουν κάποια κράτη ενώ κάποια άλλα να ξέρουν το τελείως. Και γι' αυτό ζητήσαμε γνωμοδότηση ενός καθηγητή, ο οποίος ε, κατέληξε ότι η πρόταση η νομοθετική συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και γι' αυτό θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που ήρθατε στην Επιτροπή, μας κάνατε την παρουσίαση και θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή τύχη. Καλή τύχη στην Αστριακή Προεδρία και μακάρι να έχετε πολύ θετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στα θέματα της ισότητας φύλων και της πολιτικής υπέρ της ισότητας φύλων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Colleagues, Συνάδελφοι, είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Σχέδιο έκθεσης ε, τη κυρία Πιτσέρνο για τα μέτρα για την ε, αποτροπή της ηθική και σεξουαλικής παρενόχληση στον χώρο εργασίας, δημόσιους χώρους και στον πολιτικό βίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινάμε ψηφοφορίες. Τροπολογία 48. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Πολύ ευχαριστώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Για τη 49 άρχεται η ψηφοφορία και τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41 λέει πρόεδρος υπέρ κατά αποχές «51» διορθώνει η Πρόεδρος. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 51. 51, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 52. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 56 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 58 με την προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Η συγκέντρη είναι υπέρ, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 60, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 68. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 69 και 70 μαζί ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται τροπολογία απορρίπτονται και τώρα πάμε στην 71 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται τέλος το ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για την 71 λίγη ψηφοφορία απορρίπτεται ισοπαλία βοηθάει ο έλεγχος τροπολογία 72 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικό έλεγχο και για την 72 άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 74. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβεστική τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 82. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 81. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 94 άκτη ψηφοφορία mm. τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται 95 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 96 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και εγκρίνεται. Τροπολογία 99. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. 98 τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 97. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 100. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 105 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 106 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 107. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 109 άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας και εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 14 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 115 με την προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Ποιο είναι υπέρ? Κατά αποχές εγκρίνεται. 116 σε δύο τμήματα. Ποιο... Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 117 με την προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 118. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικό έλεγχο για την συμβαστική τροπολογία 15. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16. Ποιο είναι υπέρ. <coughs> Κατά απόχε. Εγκρίνεται. Τα 127 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο ερώτημα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και αυτό. 126, ποιος είναι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 131 σε δύο τμήματα υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται και δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο της 132 μάλιστα άρχεται η ψηφοφορία για την 132 Τέλος ψηφοφορίας και απορρίπτεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 136. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 138. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 1 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 9. Υπέρ. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Αν θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Καλώς για την 9 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 11. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 με την προφορική τροπολογία του ΕΛΚ ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 με την προφορική του ΕΛΚ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 54. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 29 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 32. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 33. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται αλλά στο ελέγξουμε καλό κακού άρχεται η ψηφοφορία για την 39 τέλος ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία 38 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε το σύνολο της έκθεσης όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση άρχιτη ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ. Καλέ. Συγχαρητήρια κυρία Πίνα Πιτσένα, αλλά συγχαρητήρια και στους και ηγητές. No. ah, good, yeah. Point 12 on the agenda. Σημείο 12. Η δημοσιονομική διαδικασία του προπολογισμού. Μάλιν Μπιόρκ, ε, εισηγήτρια. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Θέλετε να ελέγξουμε τη 2. Ωραία.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 Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά αποχές. Τι θέλετε. Uh, amendment 22. It was in two parts. Yes. So. 22 ήταν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 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έκτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην τροπολογία 29, τρία τμήματα αυτής. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ,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 αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 38 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 39 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 40 υπέρ, σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν έχουμε τελική ψηφοφορία. Ευχαριστώ την συγκεκριτή Μάλιν Μπιόρκ για πολύ καλή δουλειά και τους κοιόδης εισηγητές. Ευχαριστούμε. Next. Next, next point. Ε, ε, Επόμενο σημείο 13. Πώς θα προχωρήσουμε στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον προπολογισμό για την ισότητα των φύλων. Λοιπόν, η κυρία Αγγέλικα Μίλνερ έχει ετοιμάσει το κείμενο, ψηφίζουμε. Τις τροπολογίες του ΕΛΚ κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τελική ψηφοφορία για την προφορική ερώτηση ως ετροποποίηθη, ονομαστική ψηφοφορία που ξεκινάει, πέρας, εγκρίνεται συγχαρητήρια στην κυρία Αγγέλικα Μλίνερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Now. Yeah, votes are over and now we are... Τελείωσαν οι ψηφοφορίες. To the point 14. Στο σημείο 14. Yes, point 14, just a moment. Thank you very much. Everything was okay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 She's here. She's here. Some good words from from me. Yeah. <laughs> okay. Okay. Okay. Yeah. Uh, colleagues, we now are... Συνάδελφοι, σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης. διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξέταση σχεδίου γνωμοδοτήσεως. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μαρία Ερένα, η οποία είναι εισηγήτρια για την γνωμοδότηση αυτή. No, Maria Elena. But she was here. Yes. Just a moment. Περιμένουμε λίγα λεπτά για να έρθει η συγγήτρια, η Μαρία Αρένα. Εδώ ήταν. Στην ψηφοφορία εδώ την είχαμε. Α, να τη. Συνάδελφοι, σημείο 14 της ημερησίας διατάξης. Διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση, την κυρία Μαρία Ρένα. Έχει το λόγο Μαρία. Ευχαριστώ. Είμαι λίγο αφηρημένη σήμερα. Δεν ξέρω τι τρέχει. Διακοπές, ε. Μύρισαν διακοπές. Α, εγώ δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο και λυπάμαι. Είμαι φεμινίστρια και είναι πολύ ματσό το ποδόσφαιρο και δεν βλέπω ποδόσφαιρο. Λυπάμαι κυρία Πρόεδρε που καθυστέρησα είναι σημαντικό λοιπόν στην έκθεση να μπορέσουμε να, έχουμε, να βασιστούμε στο θέμα γυναικών. Μας κατηγορούν ότι δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες όσον αφορά τη γυναίκα σε αυτό το πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε σκληρά στις διάφορες επιτροπές για να μπορέσουμε να εντάξουμε την έμφυλη διάσταση. Πιστεύω ότι στην Επιτροπή Γυναικών θα έχουμε μεγάλη ομοφωνία όσον αφορά αυτό το θέμα, διότι γνωρίζω ότι σε άλλες επιτροπές η έμφυλη προσέγγιση δεν είναι κάτι εύκολο. δεν έχω υπόψη μου τις προθεσμίες. Έχετε υπόψη τις προθεσμίες από πλευράς γραμματείας. Μπορείτε να τις κοινοποιήσετε τις προθεσμίες στα μέλη. Η αφηρημάδα μου του τέλους του έτους πριν τις διακοπές οδηγεί στο να μην έχω τις προθεσμίες. Ίσως η γραμματεία μπορεί να μας ενημερώσει δεόντως από αυτού. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μαρία Ρένα. Στου Κιώδη να δώσω το λόγο. Η κυρία Σέντροβα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Η πρόταση οδηγίας αυτή είναι σημαντική και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερε επιπτώσεις στην ισότητα των δύο φύλων. Εάν θέλετε, Μπορούμε να το χωρέσουμε και αυτό, αλλά κατά τη γνώμη μου αυτό δεν είναι απαραίτητο. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι γυναίκε είναι πιο ευάλωτε. αλλά όχι απαραίτητα να εισάγουμε συγκεκριμένε νομοθετικές διατάξεις. Η συγγήτρια είναι πολύ φιλόδοξη στις προτάσεις της. Καταλαβαίνω ότι η συνάδελφος, η κυρία Αρένα, θέλει να ενισχύσει την προστασία των εργαζομένων, Φοβάμαι όμως ότι μερικές φορές αυτό μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό και ιδιαίτερα για τις γυναίκες σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, οι πιθανές παρεκκλήσεις στο πεδίο εφαρμογής που μπορούν να υιοθετήσουν τα κράτη-μέλη. Η συγγήτρια αφαιρεί και τη μία παρέκκληση που υπάρχει. Φοβάμαι ότι αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην απασχόληση των γυναικών. Το να αφαιρέσουμε όλες τις παρεκκλήσεις ε, θα αυξήσει το διοικητικό άχθος των εργοδοτών, διότι θα πρέπει να εκδίδουν γραπτή δήλωση για όλους τους εργαζομένους, ακόμα και αυτούς που εργάζονται για πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Οι γυναίκε έχουν κυρίως τέτοιε θέσει απασχόλησης, διότι έτσι μπορούν να φροντίζουν και τα παιδιά τους και να εργάζονται με μερική απασχόληση όταν επανέρχονται στην εργασία. Ένας από τους βασικούς στόχου που θέλουμε να πετύχουμε με την οδηγία για την, τον συνδυασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου είναι οι γυναίκε να επιστρέφουν πιο γρήγορα στη δουλειά μετά την εγκυμοσύνη. Φοβάμαι λοιπόν ότι αν ο, εργοδότης πρέπει να ε, υποβάλει γραπτή δήλωση ακόμα και για εργαζόμενο που εργάζεται λίγες ώρες μόλις κάθε μήνα, θα προτιμήσουν ε, να μην προσλάβουν τέτοιους εργαζομένους, κάτι που θα επηρεάσει την ε, εξέβρεση δουλειάς που να είναι συμβατή και με τη φροντίδα των παιδιών. Όσον αφορά τις συμβάσεις μηδενικού χρόνου, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ασχολείται με το θέμα αυτό και προφανώς δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Δεν συμφωνώ λοιπόν με τη συμπερίληψη του θέματος αυτού. Επιπλέον, διαφωνώ με το ότι η συγγήτρια έχει αφαιρέσει την πιο ευνοϊκή μεταχείριση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά τις ε, συνθήκες εργασίας. Το να προστατεύσουμε τις μικροπροσθέσει επιχειρήσει από το υπερβολικό διοικητικό άχθος σημαίνει προστασία των εργαζομένων. Εάν δεν αναπτύσσονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, μπορεί να αρχίσουν ε, να χάνουν θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικές είναι οι επιχειρήσεις αυτές για την οικονομία μας με την πρόταση αυτή για τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων θα πρέπει να επιδείξουμε λογική ευελιξία. Δεν θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις ε, ε, ασυνήθιστες μορφές απασχόλησης ε, με κάθε κόστος. Θα πρέπει να τους επιτρέψουμε να αναπτυχθούν εφαρμόζοντας στην αρχή της ελάχιστης ε, προβλεψιμότητας. Ε, μάλιστα, εγώ είμαι διατεθειμένη να υποβάλω τροπολογία για περισσότερη ευελιξία. Σύμφωνα με την πρόταση, η έννοια του εργαζομένου θα βασίζεται στην ομολογία του δικαστηρίου. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα ότι κάθε κράτος μέλος έχει κάπως διαφορετικό ορισμό, κάτι που θα πρέπει να σεβαστούμε για λόγους ασφάλειας δικαίου. Είμαι λοιπόν υπέρ τροπολογίας που να στηρίζει τη, τους εθνικούς ορισμούς. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας και ελπίζω να έχουμε καλές συζητήσεις και καλό αποτέλεσμα, δηλαδή μια καλή γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια και τους Κιώδης για την σημαντική δουλειά που έχουν κάνει και για τις προτάσεις που έχουν υποβάλει. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Κάτι που δεν αναφέρθηκε, υπάρχει όμως στη γνωμοδότηση και είναι η νομική βάση. Ένας από τους στόχους της πρότασης αυτής είναι η συμμεταχείριση ανδρών και γυναικών. Η νομική βάση όμως φαίνεται μάλλον φαίνεται, ενδείκνυται να διατηρήσουμε τη νομική βάση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει να κάνει με τις ε, συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους. Κατά την εκπόνηση της πρότασης αυτής, Λάβαμε υπόψη μας το θέμα της ενσωμάτωσης της διάστασης ε, της ισότητας των δύο φύλων και θέλαμε να έχουμε μία πρόταση ε, που να προωθήσει την ισότητα των δύο φύλων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει αυτό να αποτελέσει και τη νομική βάση. Ταυτόχρονα, ο στόχος της πρότασης είναι οι ίσες ευκαιρίες κάποιες παρατηρήσεις από την μελέτη αντικτύπου για να καταλάβετε γιατί έχουμε υποβάλει την πρόταση αυτή. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες υπερεκπροσωπούνται στις μη τυπικές μορφές απασχόλησης. Επίσης, στους ανθρώπους που εργάζονται χωρίς τη θέλησή τους σε μερική απασχόληση, με συμβάσεις μηδενικού χρόνου, ή με χρόνο εργασίας 1 έως 8 ώρες την εβδομάδα. Κάτι που δεν ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογή της προηγούμενης οδηγίας. Κατόπιν έχουμε τους οικιακούς βοηθούς, όπου βλέπουμε επίσης ε, περισσότερες γυναίκες. Θέλουμε λοιπόν να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας όλων των εργαζομένων και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων ομάδων. Θέλουμε λοιπόν να στηρίξουμε τις γυναίκες και τους ανθρώπους σε επισφαλείς θέσεις εργασίας που συνήθως είναι γυναίκες. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες. Και γι' αυτό, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχουμε εξαλείψει την παρέκκληση για Όσου εργάζονται μία έως 8 ώρες την εβδομάδα. Και γι' αυτό προτείνουμε μία κατηγορία μία έως 8 ώρες το μήνα. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο ήδη έχει την εξαίρεση αυτή για τον υψηλότερο αριθμό ωρών. Μας ενδιαφέρει η εφαρμοσιμότητα από πλευράς των εργοδοτών και η προστασία των εργαζομένων σε επισφαλείς θέση εργασίας. Και όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι σημαντικό για μας να φροντίσουμε να προστατεύονται με τον κατάλληλο τρόπο και γι' αυτό εισάγουμε μια σειρά από από στοιχεία. Δεν θα έλεγα πρόταση, διότι δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε λοιπόν κάποιους πίνακες. Τα κράτη-μέλη πρέπει να καταρτίζουν αυτούς τους πίνακες και οι εργοδότες θεώρησαν ότι αυτός είναι πολύ καλός τρόπος να αντιμετωπιστεί το υψηλό διοικητικό άχθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, να υπάρχουν δηλαδή έτοιμα έντυπα για τη συμπλήρωση των στοιχείων. Ε, το πρώτο στοιχείο των επισφαλών θέσεων εργασία είναι η μη αναγνώριση. Το δικαστήριο επί 30 χρόνια δείχνει σαφώς ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκλείσουν με αυθαίρετο τρόπο ανθρώπους από την ισχύ του ευρωπαϊκού δικαίου. Και αυτό ήδη συμβαίνει. Και γι' αυτό, εάν χρησιμοποιήσουμε τους εθνικούς ορισμούς στην οδηγία αυτή, ουσιαστικά θα λέμε ψέματα στους εργοδότες και τους εργαζομένους. Θέλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα, διασφαλίζοντας και ομοιομορφία στην εφαρμογή. Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό και πολύ ευχαριστώ θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις. Για να διευκρινίσουμε και αυτό το σημείο που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό για την αποτελεσματικότητα της πρότασης και την προστασία όλων των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς και για να ολοκληρώσουμε θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Ρενά. Ευχαριστώ, όπως είπα και στην εισαγωγή. Αυτό που έχουμε να κάνουμε κυρίως είναι να πείσουμε ότι η Επιτροπή μας και η θέση των γυναικών στην πρόταση θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη. Και με εκπλήσει κάπως ε, η παρατήρηση συναδέλφου ότι δεν υπάρχει υπάρχει ιδιαιτερότητα για τις γυναίκες. Το θέμα της επισφαλούς απασχόλησης ε, αφορά κυρίως ε, και ιδιαίτερα τις γυναίκες στην Ευρώπη. Γι' αυτό και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα ενημέρωσης. Και η πρόταση αυτή στηρίζεται ακριβώς ε, στο είδος των πληροφοριών που δίνουμε στις γυναίκες. Για παράδειγμα, σήμερα έχουμε μεγάλη ανισότητα στους μισθούς Δηλαδή, για ίδια εργασία οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο από τους άντρες. Είναι δυνατόν με την πρόταση αυτή να συμπεριλάβουμε και την υποχρέωση ε, δημοσίευσης ε, των μισθών για να έχουμε περισσότερη ενημέρωση για το θέμα των μισθών και για τις μισθολογικές διακρίσεις. Γιατί μερικές φορές ε, εξηγούνται οι μισθολογικές διακρίσεις ε, από την άγνοια των γυναικών ε, για το πώς αμείβονται συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Ε, όπως εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ξέρουμε πόσο αμείβονται οι συνάδελφοι άντρες. Και σε τέτοια περίπτωση ε, εμείς όμως το γνωρίζουμε γι' αυτό και μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Αν δεν γνωρίζαμε όμως τις αμοιβέ των ανδρών συναδέλφων, μπορεί να μην διεκδικούσαμε στους μισθούς. Το ίδιο ισχύει και τους άλλους υπαλλήλους, για τους ε, διερμηνείς για παράδειγμα. Χάρη σε αυτή τη διαφάνεια των μισθών έχουμε ε, εξαλείψει τις ε, μισθολογικές διακρίσεις. Το θέμα της διαφάνειας, της ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και έδωσα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Υπάρχει ιδιαιτερότητα λοιπόν. Άκουσα το επιχείρημα που επέσε την προσοχή μας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σίγουρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητα των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Γιατί όταν μιλούμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη, μιλούμε για επιχειρήσεις που απασχολούν 200, για 250 υπαλλήλου. Αυτό όμω είναι το 90% του ευρωπαϊκού οικονομικού ιστού. Αλλά λέμε ε, να μην επιβαρύνουμε γραφειοκρατικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, δηλαδή τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους, ουσιαστικά έτσι ε, αποκλείουμε πάνω από 80% του ενεργού οικονομικού κλάδου στην Ευρώπη. Δεν συμφωνώ να εξαιρούμε 80% της οικονομίας μας από την πρόταση. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ εύστοχη σε ό,τι αφορά την ενημέρωση. Και το θέμα των πολύ μικρών επιχειρήσεων μπορούμε να το εξετάσουμε. Όταν έχουμε μια πολύ μικρή επιχείρηση να μην ε- την επιβαρύνουμε με υπερβολικό γραφειοκρατικό άγχος για την παροχή πληροφοριών. Να δούμε αν μπορούμε να βρούμε τομεακές λύσεις ε, και επιμέρους λύσεις με συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή εργοδοτών και εργαζομένων, εργοδοτών και συνδικάτων για την ενημέρωση παρόλα αυτά των εργαζομένων. Λέω ναι στην ελάφρυνση του γραφειοκρατικού άχθους για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αλλά λέω όχι στην εξαίρεση μαζικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 80 με 85% του συνολικού οικονομικού κλάδου. Δεν μπορούν να αποκλειώνται τόσο μαζικά. Ευχαριστώ Μαρία. Η τροπολογία για την κατάθεση των τροπολογιών λήγει στις 12 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Ευχαριστώ. Και περνάμε στο επόμενο σημείο, το 15 της ημερήσιας διάταξης, το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δημοσιονομικό έτος 2019. Όλα τα τμήματα. Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης της κυρίας Μάλιν Μπιέρκ. Έχεις το λόγο, Μάλιν. Uh, well, I will be very... Θα είμαι λακωνικότατη. Μόλις ψηφίσαμε τις τροπολογίες του προπολογισμού, τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις. Ευχαριστώ όλους. Σημαντικότητα τη συνεισφορά μας στην Επιτροπή Προπολογισμών. Σύμφωνα με τις γραμμές που ψηφίσαμε στα πλαίσια της γνωμοδότησης για την εντολή και θα επεξεργαστούμε το ψήφισμα που θα συνοδεύσει τον προπολογισμό αργότερα αυτό το χρόνο. Κινήθηκα όπως πριν, στα πλαίσια της εντολής. Ε, μεταφράστηκε η προσέγγιση όμως σε στοιχεία αριθμητικά που τροποποιήθηκαν και στέλνουμε ισχυρότερο μήνυμα που θέλουμε την έμφυλη διάσταση στον προπολογισμό, αντίκτυπο συνεπειών, να δούμε πού πηγαίνουν τα χρήματα. Πρέπει να επενδύσουμε στις γυναίκες, στα κορίτσια και στην ισότητα των φίλων. Είναι αρκετά σύντομη η έκθεση, θα υποβάλω και εγώ τροπολογίες. Προσβλέπω στην δική σας συνεισφορά. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρότατα προβλήματα όσον αφορά τον προϋπολογισμό για τις γυναίκες. Μείωση του χώρου, μείωση των επενδύσεων για γυναίκες και κορίτσια και μείωση του περιθωρίου κινήσεως των γυναικών στην κοινωνία είναι πραγματικότητα. Ήθελα αυτά να τα προωθήσω στα θέματα και ακόμα πιο πέρα. Με τη βοήθειά σας μπορώ να το κάνω και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ. Πιτσέρνου για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια για τη δουλειά που κάνει. Θα προσθέσω ελάχιστες σκέψεις σε αυτές που ήδη εξέφρασε η συγγήτρια. Πολλές από τις συζητηθήσεις προτεραιότητες συμπεριελήφθησαν στην γνωμοδότηση του προπολογισμού. Όμως, συμμερίζομαι αυτό που έλεγε η συγγήτρια πριν από λίγο. Πρέπει να διατηρήσουμε την προσοχή επί της ανάγκης να υπάρχει ένας προπολογισμό που σε ό,τι επίπεδα εντάσσει την έμφυλη διάσταση, κυρίως και για τα θέματα που συζητούσαμε πριν που ανέφερε η Αρενά. Ε, θα πρέπει να έχουμε καλύτερη χρήση των διευθυντικών ταμείων για να υποστηρίξουμε όλα τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών έχοντας έναν προπολογισμό που στηρίζει αυτές τις προτεραιότητες και την έμφυλη διάσταση και συμπεριλαμβάνεται στις προτεραιότητες αυτή η διάσταση του Κοινοβουλίου, αν γίνει αυτό, όλα αυτά που συζητάμε και αυτά που συζητήσαμε όσον αφορά την απασχόληση των γυναικών γίνονται αυτομάτως σημαντικές προτεραιότητες. Αυτά θεωρώ ότι είναι τα ουσιαστικά σημεία. Θα υποστηρίξω και τα άλλα σημεία βέβαια. Το αίτημα για ένα προπολογισμό ισχυρότερο που στηρίζει, και αυτή είναι η προτεραιότητα, να μην το λησμονούμε ποτέ, κυρίως αυτή την Επιτροπή, να υποστηρίζει την μάχη κατά της εμφυλής βίας. Ψηφίσαμε πριν από λίγο την έκθεση που αφορούσε την καταπολέμηση όλων των βιοπραγιών κατά των γυναικών. Βέβαια, τι σημαίνει αυτό νομικά και δικαστικά πρέπει να αναλυθεί και χρειάζονται όμως και οικονομικά μέσα. Οικονομικά μέσα δεν είναι κενά στοιχεία, δεν είναι στήρα νούμερα, είναι πολύ σημαντικά μέσα μέσω των οποίων υλοποιούμε τις πολιτικές προτεραιότητες που θέτουμε. Εκεί λοιπόν η καταπολέμηση της έμφυλης βίας πρέπει να παραμείνει κατά την άποψή μου, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είναι άποψη αυτής της Επιτροπής και να είναι προτεραιότητα θεμελιώδη. θεμελιώδης. Να εφαρμοστεί και να κυρωθεί η σύμβαση το, της και όλα τα μέσα που εξυπηρετούν στο να δίνουν ασφάλεια στις γυναίκες και καταπολεμούν ε, κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών. Αυτά είναι τα θεμελιώδη, Πρόεδρε. Θα επιφυλαχθώ όμω να συνεργαστώ με την εισηγήτρια όπως κάναμε και πριν για περαιτέρω διευκρινήσει και συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Να πω ότι είναι χαρά να συνεργαστούμε για τον προπολογισμό. Εντοπίζουμε τους ίδιους κινδύνους και ανάγκες και είμαστε έτοιμες να λάβουμε τολμηρές αποφάσεις για τα χρήματα που χρειάζονται. Το κάναμε αυτό και στα αριθμητικά στοιχεία. Και τώρα όσον αφορά τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα, κατά πολέμηση της βίας κατά των γυναικών, το μήνυμα πρέπει να είναι ισχυρότατο που θα αποστείλουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών. Πρέπει να το καταλάβουμε σαν αυτού του συναδέλφου στο Κοινοβούλιο. Αν δεν προσέξουμε τα συμφέροντα των γυναικών και τα, τη χρηματοδότηση των δικαιωμάτων των γυναικών, κανεί άλλο δεν το κάνει. Έχουμε σημαντικότατο καθήκον σε αυτή την Επιτροπή να εκτελέσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών 13 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι. Ήταν το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Να σας υπενθυμίσω ότι 3 Σεπτεμβρίου επόμενη συνεδρίαση, μετά τις θερινές διακοπές, το απόγευμα, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν τελευταία συνεδρίαση πριν τις θερινές διακοπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή δουλειά που κάναμε μαζί. Σαν μεγάλη οικογένεια εργαστήκαμε μαζί. Ευχαριστώ όλους τους ευρωβουλευτές, ευχαριστώ τους διερμηνείς, ευχαριστώ όλους τους βοηθούς, τη γραμματεία. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι να περάσετε πολύ περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές σας. Καλή ανάπαυση. Θα τα ξαναπούμε, θα ξαναειδωθούμε στις 3 Σεπτεμβρίου. Μην το ξεχνάτε. Ευχαριστώ πολύ. Από τις 12 και κλεισμένων των θυρών συντονιστές. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Μικρό διάλειμμα.